Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seat? Καλησπέρα σας, σας παρακαλώ να καθίσετε. I open the meeting of the Committee for Regional Development. Ξεκινάμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη, την οποία θα εγκρίνουμε. Θα ήθελα να σας προτείνω και μια αλλαγή. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε μια κατεξουσιοδότηση πράξη ε, την οποία ε, σας μοίρασα πολύ πρόσφατα ως σχέδιο κειμένου το Δεκέμβριο του 2014. Αναφέρομαι λοιπόν στο σημείο αυτό και να σας πω πως το τελικό σχέδιο της κατεξουσιοδότησης πράξης ε, σας μοιράστηκε στις 29 Απριλίου του 2015. Είναι τεχνικά θέματα για τα ΣΒΙΤ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει ή όχι κατά την Ολομέλεια της, του Ιουνίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας δώσει λοιπόν τώρα, ε, θα μας κάνει μια σύντομη ε, παρουσίαση του τι βρίσκεται σε αυτή την καταξιοδότηση πράξη αύριο ε, πριν λήξει η συνεδρίαση και μέχρι τις 11 Μαΐου μπορείτε να στείλετε σχόλια ή να ζητήσετε μια παράταση αν δέχεστε λοιπόν αυτή την προσθήκη στην ημερήσια διάταξη, δηλαδή το ότι προσθέτουμε μία, ε, ένα επιπλέον σημείο για την αυριανή συνάντηση, επαναλαμβάνω μία σύντομη παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατεξουσιοδότηση πράξη, λοιπόν, αν το δέχεστε σας προτείνω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Βαντίστερλο. Ευχαριστώ πολύ. Φανταζόμαστε ότι μπορεί να έρθει και η Επίτροπος, γιατί ε, χρειάζεται να μας δώσει κάποιε απαντήσεις το συντομότερο δυνατόν. Οπότε φανταζόμουν πω θα είναι εδώ τώρα, μια που είναι ήδη Μάιο. Πείτε μου όμως, τι θα κάνει, θα έρθει, θα έχει χρόνο να απαντήσει ερωτήσει μας. Για την τελευταία φορά θυμόσαστε, χρειάστηκε να φύγει τρέχοντα. Και τελικά δεν απαντήθηκαν οι ερωτήσει μα. Έχετε κανονίσει κάτι, έχουμε λοιπόν αρκετό χρόνο για όταν θα μας επισκεφθεί. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Είχα σκοπό να σας πληροφορήσω ε, κατά την συνάντηση των συντονιστών, γιατί εκεί θα ληφθεί η απόφαση, πως πρόκειται να καλέσουμε εδώ την Επίτροπο και θα το ανακοινώσω τώρα και στα μέλη. Ε, να σας πω πως η Επίτροπος μας υποσχέθηκε πως θα έρθει στη συνεδρίασή μας τον Ιούνιο. Σίγουρα έχει προγραμματιστεί. Θα έρθει λοιπόν σε μια συνάντηση που θα κάνει η Επιτροπή μας τον Ιούνιο. Τώρα για το θέμα του χρόνου που θα διατηθεί, θα προσπαθήσουμε να τη διαθέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για να έχει ε, τη δυνατότητα να απαντήσει σε όλα μας τα ερωτήματα και σε ερωτήσεις από την προηγούμενη φορά και βέβαια έχουμε νέα θέματα, νέες ερωτήσεις και αυτά πρέπει να συζητηθούν. Θα έρθει λοιπόν τον Ιούνιο. Εγκρίνεται λοιπόν η σε διάταξη. Πολύ ωραία. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο. Έγκριση των πρακτικών. Έχουμε το σχέδιο πρακτικών για τη συνεδρία στις 26 Μαρτίου. Επαναλαμβάνω, 26 Μαρτίου. Λυπάμαι. Λυπάμαι, δεν συνεδριάσαμε τον Απρίλιο, γι' αυτό έχουμε εδώ τα πρακτικά από την συνεδρίαση της 26 της Μαρτίου. Τα έχετε στο φάκελό σας. Αυτό που προτείνω είναι, αν δεν έχετε αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, να, θεωρούμε πως, ε- να θεωρήσουμε με συγχωρείτε πως εγκρίνονται. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Δύο ανακοινώσεις έχω να σας κάνω. Αύριο έχουμε αρκετές ψηφοφορίες. Στις 10 το πρωί. Παρακαλώ να είστε στην ώρα σας. Και να φέρετε μαζί και την κάρτα για να μπορείτε να ψηφίσετε. Γιατί θα γίνουν ονομαστικές ψηφοφορίες αύριο. Δεύτερη ανακοίνωση. Αύριο στις 2 παρατέταρτο θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, 1 και 45 λοιπόν, θα μας ενημερώσουν οι εκπρόσωποι της DG Regio για το πρώτο θέμα που έχει συνημερίσει η διάταξη η ομάδα εργασίας. Αυτά από εμένα. Ίσως Ίσως ε, δεν έχω καταλάβει κάτι, αλλά έχουμε και μια αργία τώρα το Μάιο στις Βρυξέλλες, έτσι δεν είναι. 25 Μαΐου είναι αργία. Είπα στις 2 παρατέταρτο αύριο. 1 και 45 αύριο. Αυτό, αύριο. Θα γίνει συνεδρίαση στην ομάδα εργασίας, τη ομάδα εργασίας εδώ αλλά όχι σε αυτή την αίθουσα, στην άλλη. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μου. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Το σχέδιο έκθεσης για τις κατευθυντήριες γραμμές Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 23 του ε, κανονισμού για τις κοινέ διατάξεις. Το άρθρο αυτό δημιουργούμε το μηχανισμό για να σχετίσουμε τη στήριξη από τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαστροτικά Ταμεία με την χρηστή διακυβέρνηση. Τον Ιούλιο πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία ανακοίνωση για το πρώτο τμήμα αυτού του άρθρου, παραγράφος λοιπόν 1 με 8, που περιγράφουν τις διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να αναπρογραμματίσουν ένα τμήμα των κονδυλίων που λαμβάνουν. Ο κύριος Λόπες θα μας παρουσιάσει σήμερα το σχέδιο έκθεσης το οποίο μας έχει ήδη ε, παρουσιάσει προκαταρκτικά τον προηγούμενο μήνα. Οι τροπολογίες παρακαλώ να υποβληθούν μέχρι το μεσημέρι της 3ης 19 Μαΐου. Noon Tuesday 19th of May. Λοιπόν, μέχρι το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι, στις 19 Μαΐου, ημέρα Τρίτη, και θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο την έκθεση αυτή. Έχουμε εδώ τον εισηγητή, κύριε Λόπες, έχουμε τους σκιώδεις εισηγητές και έχουμε και τον κύριο Ζωάζ, που είναι εκπρόσωπος, αντιπρόεδρος μάλλον της Επιτροπής Περιφερειών, ο οποίος επίσης θα μας κάνει μια παρουσίαση της, δική τους, ε, της δικής τους αφού κάνουμε και εμείς τη δική μας συζήτηση. Κύριε Λόπες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως η πλειοψηφία εδώ πιστεύει όπως και εγώ πως η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να ζητήσει μια ισόρροπη και δημοκρατική ε, εφαρμογή της αρχής ερεσιμότητας όπως θα έχουμε στο άρθρο 23 του Κανονισμού για τις Κοινές Διατάξεις των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Αυτό είναι ο στόχος της ε, έκθεσης που θα σας παρουσιάσω σήμερα. Και με το στόχο αυτό, ως κονδικό σημείο του κειμένου, συνδέεται η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με όλη τη διαδικασία αναπρογραμματισμού ή αναστολής ε, της χορήγησης ε, ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων σύμφωνα με τόσα θεσπίζει το άρθρο 23. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περίπτωση που έχουμε επαναπρογραμματισμό ή αναστολή πληρωμής κονδυλίων είναι το βασικό στοιχείο που εγγυάται την δημοκρατική, ισόρροπη, διάφανη και ευέλικτη εφαρμογή της μακροοικονομικής αρισιμότητας. Αυτή η εφαρμογή θα πρέπει να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις αρχές της πολύπλευρης ε, χρηστής διακυβέρνησης με σεβασμό της αναλογικότητας και της επικουρικότητας για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στα κράτη-μέλη, όπως επίσης και των περιφερειών που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικές δυσκολίες πραγματικές και όπου τα ευρωπαϊκά κονδύλια και ταμεία... αποτελούν μεγάλο τμήμα των προπολογισμών τους. Αυτό είναι στις παραγράφους 12, 15 και 17. Είδαμε με την ευκαιρία αυτής της τόσο δύσκολης κρίσης ε, που αντιμετωπίζουμε, πως αυτά ακριβώς τα ευρωπαϊκά ταμεία στην πράξη ήταν η μοναδική επένδυση που λαμβάνει η χώρα σε πολλές περιοχές και περιφέρειες της Ευρώπης. Το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσουν ένα διαρθρωμένο, δομημένο διάλογο που θα εξασφαλίσει πως θα υπάρχει διαθεσμική, διαθεσμικό συντονισμός και η απαραίτητη ροή πληροφοριών για όλες τις διαδικασίες σύμφωνα με τα όσα θεσπίζει το 23. Το Κοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει τουλάχιστον να ενημερώνεται αμέσως, αυτό είναι το ελάχιστο, για οποιοδήποτε αίτημα αναπρογραμματισμού ή αναστολής πληρωμών. Έτσι έστε να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη θέση του εν ευθέτω χρόνο και με τον τρόπο που θα επιτρέψει να ληφθεί υπόψη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, από την οποία απαιτούμε να α, κάνει έναν απολογισμό και μια λογοδοσία για ό,τι δράση αναλαμβάνει στις περιπτώσεις αυτές. Για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περίπτωση επαναπρογραμματισμού και αναστολής, παράγραφη 24 και κάτω, Νομίζω ότι αυτό θα μείνει σε κρεμότητα μέχρι τη συζήτηση και την ενδεχόμενη πιο συγκεκριμένη διατύπωση που θα βασιστεί στις τροπολογίες που θα υποβληθούν και στους συμβιβασμούς στους οποίους θα πετύχουμε τις επόμενες εβδομάδες με τις υπόλοιπες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί πιστεύω πως το θέμα αυτό απαιτεί τη μεγαλύτερη δυνατόν συνένεση από όλες τις πολιτικές ομάδες. Εκτός από το σημείο αυτό πρέπει να σου πω πως θέλουμε μια έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει επιπλέον ε, επιπλέον στοιχεία για την επίπτωση των μακροοικονομικών αυτών ε, μεγεθών στην περιφερειακή ανάπτυξη και πώς συνδέεται η ευρωπαϊκή ε, πολιτική, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ε, τη χρηστή διακυβέρνηση στα ευρωπαϊκά κράτη, με συγκεκριμένες συνθήκες και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με συστάσεις ανακράτος, σύμφωνα ε, με τα όσα έχουν αυξηθεί στο Συμβούλιο. Ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού τα κράτη-μέλη, να κάνει μια ανάλυση όλων των εναλλακτικών λύσεων που είναι διαθέσιμες και οι οποίες είναι, που διαφέρουν κατά τη από το άρθρο 23 παράγραφος 10 και θα θέλαμε να μας ξεκαθαρίσει με πιο συγκεκριμένο τρόπο θα λαμβάνει υπόψη τις οριζόντιες αρχές του κανονισμού σε ε, διαβούλευση και σε ε, συζήτηση με τα κράτη-μέλη της περιφερειακής και τοπικής επίπτωσης των μέτρων που θα ληφθούν στα πλαίσια του άθρου για το οποίο συζητάμε. στην έκθεση που αναφέρεται στις επιπτώσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το 23 όταν έχουμε συγκεκριμένα ποσά ε, και συγκεκριμένα μέτρα πώς αυτό επηρέασε και την ανταγωνιστικότητα των ταμείων αλλά και την ανάπτυξη γενικότερα. Αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία της έκθεσης που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά. Όλα αυτά από μια οπτική γωνία η οποία ε, αντιμετωπίζει με κριτικό πνεύμα την μακροοικονομική ρεσιμότητα ε, και σύμφωνα με τόσα διαπιστώσαμε στη συζήτηση που κάναμε κατά τη διάρκεια της πρώτης ανταλλαγής απόψεων για το θέμα αυτό. Πιστεύω πως το κείμενο αυτό είναι ισορροπημένο. Και επειδή είναι αδύνατον να τροποποιήσουμε ή να διαγράψουμε το άρθρο 23 θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια εφαρμογή η οποία θα είναι όσο δυνατόν πιο δίκαιη, όσο δυνατόν πιο δημοκρατική. Παρόλο που δεχόμαστε τις σκληρές επικρίσεις ε, που έχουν απευθυνθεί για τη μακροαιρεσιμότητα, για παράδειγμα από την Επιτροπή Περιφερειών. Και όπως είπε και η Πρόεδρός μας, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τα όσα θα μας πει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Περιφερειών εδώ. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να συγχαρούμε αλλήλους για την πολύ συνετή προσέγγιση της Επιτροπής και για το στόχο αυτής να μειώσει στο μέγιστο και τον επαναπρογραμματισμό και την αναστολή πληρωμών. Γιατί τα όσα συμφωνήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις συγκεκριμένες συστάσεις κράτος και τις συστάσεις που σχετίζονται με τα θέματα που αφορούν που έχει απευθύνει το Συμβούλιο. Κάποια έμειναν στα χαρτιά. Άρα θα πρέπει μέσω τροπολογιών να δούμε τη δυνατότητα οι αναστολές και επαναπρογραμματισμός που αναφέρονται σε σχέση με την μακροοικονομική αιρεσιμότητα να αποτελέσουν και μια, ένα, τελευταίο, καταφύγιο στο οποίο θα στραφούμε όταν δεν μπορούμε με τα δικά μας μέσα να βελτιώσουμε την κατάσταση και χωρίς να θίγονται ε, επουδενή ε, οι στόχοι της πολιτικής συνοχής. Είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε σχόλιο, σε οποιαδήποτε πρόταση και θα ήθελα ο διάλογος μεταξύ μας να βασιστεί στις τροπολογίες οι οποίες θα υποληθούν από τώρα μέχρι και την ημέρα που θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λόπες. Θα δώσω τώρα το λόγο στους ε, σκιώδης Κύριε Πότσακ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή διότι μας παρουσίασε το κείμενο της έκθεσής του. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπες παρουσίασε μια έκθεση έκθεση την οποία θεωρώ ε, ποιοτική και σημαντική. Και αυτό είναι εξαιρετικό διότι ευθυγραμμίζεται και με την θέση του Κοινοβουλίου για το άρθρο 23 και τις ε, ε, διάφορες περιπλοκές του. Πρόκειται για ένα άρθρο το οποίο δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί και θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως ε, να πάρει μια νέα απόφαση, μια νέα εκτελεστική απόφαση και ενδεχομένως να αποφασίσει ανέρεση, διότι όχι διότι υπάρχει ρήξη ε, κάποιων διατάξεων, η παράβαση κάποιων διατάξεων, αλλά λόγω γενικότερης εμπορικής ε, καταστάσεως ελήφθησαν υπόψη ε, πολλά στοιχεία για την έκθεση αυτή και ελήφθησαν σαφώς υπόψη από τον εισηγητή και τα σχόλια των συναδέλφων στη συνεδρίαση του Μαρτίου. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να πω ότι η πρόταση είναι πολύ σε ποιότητος ε, και απλώς μπορούμε να προσθέσουμε κάποια πράγματα, όπως ε, ας πούμε στο σημείο 8 ε, εκεί που μιλάμε για εταιρικέ σχέσεις και συμφωνίες. Στο σημείο αυτό πιστεύω ότι οι συμφωνίες αυτές ε, μπορούν να ε, εκεί μπορούν να προσθεθούν λέω κάποια, κάποια άλλα εργαλεία ή κάποια άλλα στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν στην Κομισιόν να ε, κάνει κάτι όσον αφορά προγράμματα τα οποία δεν ευθυγραμμίζονται με κάποιες προϋποθέσεις και κάποια υφιστάμενα προγράμματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν όπου χρειάζεται επαναπρογραμματισμός ε, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό θα μπορούμε να το δεχτούμε μονάχα σε περίπτωση εξαιρετικών περιπτώσεων. Ε, στο 11 υπερβολική ε, γραφειοκρατικό ε, βάρος. Ε, όσον αφορά κάποιες ε, καθυστερήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα. Κοιτάξτε, στην ουσία εδώ έχουμε κάποιες περιπτώσεις όπου ε, προκαλούν καθυστερήσεις. Τώρα, εάν επαναπρογραμματίσουμε ε, ε, περιπτώσεις ειδικά επί των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεγαλύτερο βάρος, τότε θα επαπειληθεί κατά κάποιο τρόπο η ίδια η πολιτική συνοχής. Σημείο 17 ε, όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας. Να μην λησμονούμε ότι εάν δεν αναλάβουν τις δεσμεύσεις τους και δεν τις υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη, ε, ίσως γιατί δεν έχουν αρκετή πειθαρχία αλλά και για άλλους λόγους, ενδεχομένως γιατί δεν μπορούν ας πούμε, να ελέγξουν κάποιες ε, φυσικές καταστροφές. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην έκθεση. Σημείο 19. Παροχή πληροφοριών. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να τροποποιηθεί λίγο, κυρίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, ε, όσον αφορά την αναφορά κάποιων ε, υπηρεσιών ενωσιακών που έχουν πρόσβαση στην ε, πληροφόρηση και να πούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ε, πρόσβαση στην πληροφόρηση και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά ε, στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα το σημείο 24 ε, έως 28 της εκθέσεως ρόλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι καλύτερα θα ήταν να αναφερθούμε και στην Επιτροπή μας, δηλαδή στην Επιτροπή Περιφερειακών ε, Υποθέσεων και ενδεχομένως και την Επιτροπή των Περιφερειών, γιατί όχι. Η πρόταση είναι καλή. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπλανκό Λόπες. Χαίρομαι που συνεργαστήκαμε και επομένως είμαι πολύ ευτυχής με το σχέδιο της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ θα δώσω το λόγο στην κυρία Τόμασιτς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτή την εξαιρετική έκθεση που μας δίνει κάποια, κάποιες πολύ χρήσιμες συστάσεις για το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης. Επίσης, τονίζεται ότι οι αποφάσεις για αναπρογραμματισμό ή αναστολή πληρωμών του άρθρου 23 πρέπει να είναι πλήρως ιδιολογημένε για να υπάρχει διαφάνεια και έγκαιρη αναθεώρηση. Η πολιτική συνοχή και οι σχετικές επενδύσεις από το 2014 στο 2020 θα χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν οι πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη-μέλη και που είναι ευθυγραμμισμένες με τις ολοκληρωμένες κατευθύνες γραμμές και τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης. Ο βασικός στόχος παραμένει η εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου και βέβαια το να αποφεύγονται πολιτικές οι οποίες δεν είναι βιώσιμες. Τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία έχουν μεγάλη σημασία για να έχουμε επενδύσεις στις ε, περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό η Κομισιόν πρέπει να εφαρμόσει το άρθρο 23 σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση στις εν λόγω χώρες και περιφέρειες. Οι περιφέρειες αυτές αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικές δυσκολίες και τα επενδυτικά ταμεία είναι σημαντικό κομμάτι των συνολικών επενδύσεων. Ο συχνός αναπρογραμματισμός μπορεί να επηρεάσει την προβλεψιμότητα και έτσι μπορεί να κινδυνεύσει η σταθερότητα των συμφωνιών εταιρική σχέση και βεβαίω να έχουμε και άδικε κυρώσει για τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ, οι οποίε παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία τη Ένωση και είναι 33% των δημοσίων κονδυλίων. Απευθύνομαι άρα προ την Κομισιόν και τη ζητώ να κάνει την απαραίτητη αξιολόγηση για τον αντίκτυπο των μέτρων του άρθρου 23 σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Σα ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Φαν Μίλτενμπουργκ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος του κυρίου Όλι Ρεν, ο οποίος εξελέγει στην Φιλανδία. Όσον αφορά το σχέδιο έκθεσης θα ήθελα να τονίσω κάποιες από τις προτεραιότητες της ΑΛΔΕ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ειδικά σε σχέση με το άρθρο 23. Βεβαίως ως Άλντε θεωρούμε πως η σωστή ε, οικονομική διακυβέρνηση και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων δεν είναι κάτι αντίθετο. Μπορούν να ισχύσουν παράλληλα. Ταυτόχρονα θέλουμε να ισχύσει το άρθρο 23 και να εφαρμοστεί με τρόπο που δεν θα διακινδυνεύει η εφαρμογή της πολιτικής ε, συνοχής, να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για τους πιθανούς ετούντες ε, ή δικαιούχους των διαρθρωτικών ταμείων στο παρελθόν ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για έναν κανονισμό κοινών διατάξεων, ειδικά σε σχέση με την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Ήταν διχασμένο το Συμβούλιο, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις εντός της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε, τελικά καταλήξαμε σε έναν συμβιβασμό που βεβαίω απέχει αυτό να είναι τέλειος, αλλά πάντα αναζητούμε μια ισορροπία. Αν δούμε τώρα την έκθεση, ε, είμαστε αρκετά επικριτικοί. Θεωρούμε πως το άρθρο 23 για τη μακροοικονομική αρισιμότητα είναι αναγκαίο και βεβαίως ε, το είπα και στην, σε προηγούμενη συνεδρίασή μας ότι αυτά θα φανούν στην πράξη. Αλλά εάν δούμε την έκθεση σήμερα και δούμε το άρθρο, την παράγραφο 14 όπου αναφέρεται πως εμείς ως ε, Επιτροπή Ρέτζι δεν δεχόμαστε την ανικανότητα αυτή να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα σε εθνικό επίπεδο να καταλήγει σε ε, τιμωρία αρχών που είναι κάτω από το εθνικό επίπεδο. Μα αυτή είναι η ουσία της αρεσιμότητας, είτε μας αρέσει είτε όχι, αν σε ένα κράτος μέλος δεν υπάρχει χρηστή διοίκηση και εκεί πέρα συμφωνώ το άρθρο 23 θα εφαρμοστεί ως τελευταία λύση, όχι κάτι το οποίο θα κάνει εύκολα η Κομισιόν, αλλά η συνέπεια θα είναι ότι αρχές κάτω των εθνικών θα υποστούν τις οικονομικές συνέπειες στις δυνατότητες τους να κάνουν κάποιες επενδύσεις. Θα δούμε λοιπόν κάποιες τροπολογίες που είναι σύμφωνες με την προηγούμενη θέση της ομάδας μας και θα τη στείλουμε στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Η κυρία Μαρτίνα Άντρεσον δεν είναι εδώ, από ό,τι βλέπω. Όχι, δεν είναι εδώ. Επομένως συνεχίζουμε με την κυρία Πάνα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ πρέπει ε, να σας πω γιατί ο, ο, ο κανονικός ε, ε σκιώδης ε, δεν είναι εδώ. Εν πάση περιπτώσει οι ε, πράσινοι είναι κατά της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας γιατί πιστεύουν ότι είναι ακριβό και ανώφελο εργαλείο το οποίο περισσότερο βλαβερό θα αποβεί παρά ωφέλιμο. Παρόλα αυτά ο εισηγητής της έκθεσης αυτής πρέπει να είναι περήφανος γιατί έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά με, πολύ υψηλής ποιότητος ε, εξισορρόπησε με λογικό και κανό τρόπο ε, την ε, μακροοικονομική αιρεσιμότητα με την ανάγκη ομαλής εφαρμογής ε, των ε, προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή βάση συζήτησης. Βεβαίως εμείς έχουμε κάποιες ε, προτάσεις διατύπωσης, ας πούμε θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμιστεί ακόμα περισσότερο ότι η προσφυγή στην ερεσιμότητα αυτή θα είναι η τελευταία δυνατότητα, ούλτιμα ράσιο. Επίσης θα πρέπει να γίνει ε, σαφής αναφορά στο βάρος της απόδειξης ε, και ε, κάποια άλλα στοιχεία. Επομένως, ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει την καλή συνεργασία που είχε μέχρι τώρα ο εισηγητής με τους εσκιώδεις και θα καταφέρουμε να βρούμε συμφωνία και επί των σημείων που ανέφερα με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Συγχαρητήρια κύριε εισηγητά για την ποιότητα της έκθεσής σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεμάτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι τον συνάδελφο για την ε, εργασία του. Αναφέρεται σε ένα θέμα ιδιαίτερος ε, αμφισβητούμενο, δηλαδή αυτό της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Εγώ στο ξεκίνημα ήμουν πάρα πολύ ε, περίεργη να δω προς ποια κατεύθυνση θα πήγαιναν τα σχόλια του συναδέλφου. Το διάβασα λοιπόν όλα πολύ προφτικά. Επομένως αυτό το άρθρο 23 φαίνεται πλέον σαφώς ότι απασχολεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις και επομένως ε, χαίρομαι γιατί ο ε, εισηγητής κάνει έκκληση στα σημεία 15 και 17 ε, στην επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Στο σημείο 14 αναφέρεται στην αρχή σύμφωνα με την οποία ναι, η αδυναμία λύσης των μακροοικονομικών προβλημάτων σε εθνικό επίπεδο προκαλεί προβλήματα σε επίπεδο περιφερειών και επομένως αποτελεί πρόσκομα σημαντικό για την ολοκλήρωση της περιφερειακής πολιτικής ο ρόλος τώρα των τοπικών και περιφερειακών αρχών που δεν ευθύνονται για τα βάρη και τις αδικίες σε επίπεδο ε, κεντρικών κυβερνήσεων ε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Ε, αναγνωρίζει ότι η αύξηση του χρέους ε, προέρχεται κυρίως από τις δράσεις της κεντρικής κυβέρνησης και επομένως άδικο θα ήταν ε, να τιμωρηθούν τοπικές και περιφερειακές αρχές για κάτι που δεν οφείλεται σε αυτές. Λέμε ότι ενδεχομένως θα υπάρξει επαναπρογραμματισμός από πλευρά της Κομισιόν, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο το που συνδέεται με την αλλαγή διακυβέρνησης, ε, κίνδυνο λέω για την κοινωνική συνοχή. Συμφωνώ πάντως με τους περισσότερους συναδέλφους ότι το γεγονός ε, ότι στις κατευθυντήριες γραμμές δεν αναφέρεται ο ρόλος του Κοινοβουλίου ε, σε, στην περίπτωση του παλαιού άρθρου 23 θα πρέπει οπωσδήποτε αρνητικά να υπογραμμιστεί. Όσον αφορά τώρα την έκθεση του συναδέλφου, η γενική μου κρίση είναι ότι πρόκειται για εξαιρετική έκθεση. Ε, θα έλεγα ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ανάγκη ε, να καταγραφεί και σε τούτη την ε, έκθεση η αναφορά της ρήτρα επενδύσεων. Δηλαδή ενδεχομένως να βγουν από τον υπολογισμό του κρατικού ελλείμματος διάφορες επενδύσεις οι οποίες αφορούν τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο κυρίως μέσω της Creating Europe. Αυτά είχαν να μας πούν λοιπόν οι σκιώδεις εισηγητές. Να ακούσουμε και τον κύριο Μπουστινάρου που έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Μπλανκό Λόπες, για μια πραγματικά ένα πολύ πετυχημένο σχέδιο και πολλές σοφές ιδέες ε, που ακούστηκαν από τους σκιώδες συζητητές είμαι σίγουρος πως θα τις εντάξει και θα κάνει το ίδιο με αυτά που έκανε η Επιτροπή η δική μας πέρσι όταν τελειώναμε τη διαπραγμάτευση όχι πέρσι με συγχωρείτε το 2013 και ήμασταν τόσο πετυχημένοι. Το ουσιαστικό τμήμα εδώ είναι πως γίνεται μια ρητή αναφορά σε αναστολή που αποτελεί το μέτρο, το, πραγματικά το τελευταίο μέτρο που μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ίστατο με απόλυτη διαφάνεια και με την απόλυτη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της Επιτροπής μας. Αυτό είναι ουσιαστικό, γιατί και οι δύο συνεισηγητές με τον τρόπο αυτό ε, σχεδίασαν τους κανόνες αυτούς για την μακροοικονομική αρισιμότητα. Και εδώ το πνεύμα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε είναι το εξή. Να μην γίνεται αυτή η αναστολή, γιατί όταν επιβάλλεται αυτή η κύρωση στι κεντρικέ κυβερνήσει για μακροοικονομικούς λόγους, τελικά το λογαριασμό τον πληρώνουν οι περιφέρειες. Και η πολιτική συνοχής έλεγε να μην υποστούν ποτέ ε, τέτοιου είδους ε, οι περιφέρειες. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει δύο και τρεις φορές οποιαδήποτε ενδεχόμενη αναστολή για να μην υπάρχει σόρευση και να μην έχουμε αυτό το σορευτικό κανόνα επιπτώσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε αναστολή. Πρόληψη τη σωστή χρονική στιγμή και ας μην χρονίζουν τα προβλήματα των διαχειριστικών αρχών σε κεντρικό επίπεδο γιατί ξέρετε πως η πολλή επιμονή είναι έργο του σατανά. Θα πρέπει λοιπόν και το θεσμικό και το διοικητικό πλαίσιο των διαχειριστικών αρχών να βελτιωθεί, των κεντρικών και των ε, περιφερειακών παικτών να βελτιωθεί, γιατί για καλύτερες δαπάνες, για αποφυγή των λαθών και των σφαλμάτων που σωρεύονται και τελικά μπορεί να οδηγήσουν σε αναστολή, ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε, επαναλαμβάνω, είναι το θεσμικό και διοικητικό δυναμικό που θα εξασφαλίσει πως από το σχεδιασμό του έργου και μέχρι την εφαρμογή αυτού θα είμαστε αποτελεσματικοί, θα έχουμε θετικές επιπτώσεις και αντίκτυπο και όλες οι προϋποθέσεις θα είναι εκεί έτσι ώστε να συνεχιστεί επιτυχώς αυτό το έργο. Και μόνο σε λίγες περιπτώσεις θα προχωρήσουμε σε αναστολή πληρωμών. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και πάλι για το σχέδιο αυτό κειμένου και σίγουρα θα σας βοηθήσω όσο μπορώ και εγώ και οι συνάδελφοι για να είναι καλή η έκθεση στο τέλος και θα βοηθήσει τελικά αυτή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κυρία Μελέτιτς. Ε, I like Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να τονίσω πως η ορθή η χρηστή οικονομική διοίκηση είναι η προϋπόθεση νομίζω για την επιτυχημένη πολιτική συνοχή και δεν μπορούμε να βλέπουμε ξεχωριστά την κεντρική από την περιφερειακή κυβέρνηση γιατί τελικά εξίσου συμμετέχουν στο δημόσιο χρέος. Πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη τη σημασία της ορθής ε, ...η οικονομικής διακυβέρνησης και πώς θα γίνει αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να πω σε σχέση με αυτή την έκθεση είναι το σημείο 8 στις ε, γενικές αυτές ε, σκέψεις. Ναι, υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα μια πάρα πολύ σημαντική τέτοια σκέψη στην οποία ο συγητής λέει πως οι συμφωνίες και τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχουν λάβει υπόψη τις σχετικές συστάσεις αναχώρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βασιζόμενοι σε αυτό λέτε στα υπόλοιπα μέρη της έκθεσης πως δεν θα πρέπει να γίνει επαναπρογραμματισμός γιατί έχουμε λάβει υπόψη τις συστάσεις, ε, τις εταιρικές ε, συμφωνίες ε, λοιπά Το ερώτημά μου όμως είναι το εξής εφαρμόζεται αυτό στην πράξη γιατί εγώ είδα κάποια επιχειρησιακά προγράμματα και συμφωνίες εταιρική σχέσης και πραγματικά δεν μπορούσα να βρω διασυνδέσεις με τις συστάσεις αναχώρα και πώς σκοπεύουν οι χώρες να χρηματοδοτήσουν τις συστάσεις που γίνονται μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων και ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες σχετίζονται με τις συστάσεις αναχώρα. Οπότε, ίσως εμείς ως Επιτροπή θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την ε, Κομισιόν να κάνει μια ανάλυση και να μας εξηγήσει πώς παρακολουθούν αυτή την σύνδεση. Και αν υπάρχει αυτό, τότε πράγματι δεν πρέπει να γίνεται ένα προγραμματισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Χέτμαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε και το άρθρο 23 με τη μορφή που έχει μοιάζει αποδεκτοκά το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτό είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές και ο εισηγητής ο ίδιος το λέει αυτό στην έκθεση του. Ε, ειδικά δε οι συστάσεις κομισιών είναι λογικές και σωστές. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει η δυνατότητα διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικά όσον αφορά τον τρόπο και το εύρος των αλλαγών έτσι ώστε όλοι να μπορούν να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουν τις προτινόμενες αλλαγές. Επίσης θεωρώ πως η Κομισιόν δεν θα πρέπει να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή με έτοιμα αναπρογραμματισμού. Αν υπάρχουν λόγοι για κάτι τέτοιο, η Κομισιόν πρέπει να το πει ξεκάθαρα και να το συζητήσει με τους ενδιαφερόμενους. Τα λέει αυτά ο εισηγητής, αλλά νομίζω πως πρέπει να τονίσουμε τον ρόλο της ε, πολιτικής ε, συνοχής, ειδικά δεδομένης ε, της κρίσης από την οποία μόλις βγαίνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διαρθρωτικά ταμεία και η πολιτική συνοχής ήταν ένα είδος μαξιλάρι και βεβαίω η πολιτική συνοχής κατάφερε να αποτελέσει όπως είπαμε ένα μαξιλάρι για τις πολύ αρνητικές αυτές συνέπειες. Εάν ο μηχανισμός αυτός αναπρογραμματισμού ε, εφαρμοστεί πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι απαραίτητοι παράγοντες όπως και οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές αλλά ε, σε πάρα πολλά πράγματα στο ΑΕΠ, στην παραγωγή συνοψίζοντας λοιπόν θα ήθελα να συμφωνήσω με τον εισηγητή ότι δηλαδή εφόσον συμμετείχε μέχρι στιγμή στο Κοινοβούλιο δεν πρέπει να αποκλειστεί. Κύριε Ροϊ, έχω σημειώσει το όνομά σας, αλλά ε, επιτρέψτε μου να δώσω λόγο στον κύριο Πόλτσακ που θέλει να αντιδράσει λίγο σε αυτά τα οποία είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τσανέφ αναφέρθηκε προηγουμένως αλλά, ε, σε αυτό το θέμα, αλλά και ε, ο προηγούμενος ομιλητής αναφέρθηκε στην, ε, στην ποινικοποίηση των περιοχών. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά την χρηματοδότησή τους, οι περισσότερες περιφέρειες είναι ανεξάρτητες αλλά πρέπει να σας πω ότι στην Τσεχία ε, ένα 25% των, ε, του χρέους, του κρατικού χρέους αφορά και τις περιφέρειες. Σε πάση περιπτώσει, εάν χρησιμοποιήσει αυτά τα συσταλτικά μέτρα η Κομισιόν, τότε οπωσδήποτε ο αντίκτυπος θα είναι αρνητικός και στις ε, τοπικές και τις περιφερειακές διοικήσεις. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν κάποια στοιχεία εξισορρόπησης του προβλήματος. Δεν θα πρέπει πρέπει να θεωρούνται οι περιφέρειες ε, οι υπεύθυνε για, αυτές τις, για αυτά τα χρέη. Στην Ελλάδα, ας πούμε, φαίνεται ότι ε, η κεντρική κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει χρήματα από τις περιφέρειες και τους Δήμους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον συγητή. Αν δείτε την πολιτική συζήτηση που είχε γίνει πραγματικά αφορά την ουσία του θέματος. Πρέπει λοιπόν να, να λύσουμε σωστά και να δούμε ποια θα είναι και η πολιτική της δικής μας Επιτροπής. Ε, θα ήθελα τώρα να πω κάτι για το άρθρο 14. Ετέθη το ζήτημα της απροθυμίας ε, των ε, κρατών για να αγγίξουν αυτά τα μακροοικονομικά ζητήματα. Αν είναι θέμα ανικανότητας πρέπει να τους βοηθήσουμε, αλλά αν είναι θέμα βούλησης ή μη βούλησης ε, τότε Πρέπει να δούμε γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα και αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να ξέρω και νομίζω πως αναφέρεται πάρα πολύ σωστά στο σημείο 27 είναι όταν εμείς ως Επιτροπή λαμβάνουμε κάποια γενική εικόνα των πραγμάτων που είναι άνα χώρα και αφορά, αφορούν κάποιον αναπρογραμματισμό θα πρέπει να έχουμε ένα έγγραφο, ένα, μια έκθεση ετήσιας προόδου για τα περιφερειακά κονδύλια και του άρθρου 23. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό να ζητήσουμε κάτι τέτοιο. Αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί νομίζω πως παραγνωρίζεται τη σχέση αυτού του άρθρου σε σχέση με την πολιτική μας. Και δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό αυτό που στάω, θα μας πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω πως αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιατί είναι κάτι το οποίο συζητιέται αυτή τη στιγμή και στην Επιτροπή Οικονομικών. Τι κάνουμε, τι μπορεί να γίνει με το ε, ευρωπαϊκό εξάμεινο κτλ. Και έχουμε πάλι την ίδια την ίδια ιστορία με αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα. Ωραία είναι δηλαδή ότι στις διαπραγματεύσεις δώσαμε πάρα πολύ βάρος ε, στο προληπτικό σκέλος. Όλα τα μέτρα είναι προληπτικά. όπου κοιτάμε δηλαδή να δούμε το τι μπορούμε να επαναπρογραμματίσουμε. Και δεύτερον, όταν ερχόμαστε μετά να διορθώσουμε εκ των υστέρων έχουμε βάλει πάρα πολλά πράγματα που τελικά αποτρέπουν το να γίνει οποιαδήποτε περικοπή ή διόρθωση. Μπαίνουν μέσα νούμερα ανεργίας και διάφορα τέτοια. μια απόφαση που θα έπρεπε να είναι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά υπάρχουν, ε, όπως είπα, πάρα πολλές ε, δικλείδες ε, ασφαλείας. Οπότε αν το δει κανείς, δεν βλέπει πως δεν είναι τόσο αυτόματο. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει ως τελευταία λύση και υπάρχουν πάρα πολλοί αερόσακοι θα έλεγα. Πριν φτάσει η Επιτροπή να κόψει λεφτά από το Ταμείο Συνοχής. Αλλά εγώ θα ήθελα μια έκθεση, μια τεκμηρίωση ε, στην οποία θα μπορούμε να επανερχόμαστε. Έτσι νομίζω αυτά αναφέρονται και στο 25, 26, 27. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλα μέλη να ζητούν το λόγο και επομένως θα δώσω λόγο στον κύριο Κάρθελ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν συμφωνώ απλώς με τα όσα είπε ο εισηγητής. Θα ήθελα καταρχήν να τον συγχαρώ τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά τα προσυπογράφω γιατί για 19 χρόνια ήμουνα στην ηγεσία μιας περιφερειακής κυβέρνησης και αυτομάτως ήμουνα και μέλος Επιτροπής Περιφερειών και εκεί είχαμε επικρίνει πολύ σκληρά αυτή την μακροοικονομική ερεσιμότητα. Άρα λοιπόν, να σας πω πως είμαι απολύτως πεπισμένος πως η έκθεση αυτή βασίζεται σε πολύ σωστές βάσεις, έχει πετύχει το στόχο της και πιστεύω πως περιγράφει τέλεια το τι ακριβώς πιστεύει το Ευρωκοινοβούλιο. Άρα λοιπόν συμφωνώ απόλυτα και συντάσσομαι γιατί είναι σωστή, πάρα πολύ σωστή αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να υπάρχουν ε, άλλα μέλη της Επιτροπής που να θέλουν το λόγο. Ο κύριος Σουάς λοιπόν από την Επιτροπή Περιφερειών Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι εισηγητής για την Επιτροπή Κοτέρα της Επιτροπής Περιφερειών και μάλιστα ήταν υπό την προεδρία του συναδέλφου Βαν Κάρσελ που είχαμε εγκρίνει ομόφωνα ε, μια σχετική έκθεση. Πρώτα απ' όλα μια ε, τυπική ας πούμε παρατήρηση να συγχαρώ τον εισηγητή και για την εργασία του αλλά για την ποιότητα της συνεργασίας που είχε μαζί μας ε, και πραγματικά χαίρομαι γιατί έλαβε υπόψη του τα περισσότερα από όσα είπαμε εκτός από ένα σημείο το οποίο ανέφεραν όμως άλλοι κυρίως ο πρόεδρος Κάσελ ότι επί της ουσίας εμείς αντιτιθέμετα στην μικροοικονομική αιρεσιμότητα ε, για λόγους που ήδη εκφράστηκαν από προορίσαντες εδώ αλλά εν πάση περιπτώσει μια και τα πράγματα είναι όπως έχουν εμείς ε, ως, όπως και εσείς θα προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε την υφιστάμενη συγκεκριμένη κατάσταση. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας σε κάποια ερωτήματα και κάποια ζητήματα τα οποία αναφέρω εντάχει. Θα θέλαμε να ε, ε, αναφερθεί σαφώς ο κίνδυνος και το λέω γιατί εγώ είμαι αντιπρόεδρος μιας μεγάλης περιφέρειας, της περιφέρειας Ροδανού Άλπαιων ε, και επίσης είμαι και ε, πρόεδρος ε, της Region France, των, της Ένωσης Περιφερειών της Γαλλίας και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι έχουμε συζητήσει πολλές φορές τα θέματα αυτά. Τους είπα λοιπόν προσοχή γιατί χρειαζόμαστε σταθερότητα ε, και εν προκειμένου αυτή η μακροοικονομική αιρεσιμότητα ε, δημιουργεί έλλειψη σταθερότητας ακριβώς στη λειτουργία των περιφερειών. Δεύτερο σημείο που θέλουμε να υπογραμμιστεί και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, προσεκτικοί σε αυτό. Ο επαναπρογραμματισμός είναι ένας πραγματικός δαίμονας. Βρισκόμαστε στα μέσα περίπου του 2015. Μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού τα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία έχουν ήδη ε, αρχίσει να λειτουργούν. Ναι, πρέπει να σας πω ότι η Γαλλία η οποία είναι από τους πιο προχωρημένους παίκτες δεν έχει ξοδέψει πάνω από το 1% του προϋπολογισμού. Επομένως ο επαναπρογραμματισμός μπορεί ε, σε θεωρητικό επίπεδο να είναι κάτι ευφιές. Είμαι οικονομολόγος και βγάζω θεωρίες. Αλλά όταν δει κανείς ε, τις, ε, ε, τις αργοπορίες οι οποίες προστίθενται σε αργοπορίες, όταν δει κανείς το, ε, δημοσιονομικό βάρος θα καταλάβει τι λέω. Τρίτο, αναφέρθηκε από πολλούς ε, και το σημεριζόμαστε Μια τέτοια μακροοικονομική αιρεσιμότητα οπωσδήποτε θα πρέπει να εμπλέξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπωσδήποτε. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει τη θέση του γιατί εσείς είστε νομοθέτες και επομένως θα πρέπει να συμμετάσχετε σε αυτή τη διαδικασία που δεν μπορεί να είναι απλή γραφειοκρατική διοικητική διαδικασία. Ε, λέω δε ότι σε ε, πολλές ε, περιπτώσεις, σε πολλές ε, χώρες μπορεί να υπάρχει περιφέρεια η οποία να κυβερνάται από ένα πολιτικό κόμμα το οποίο είναι αντίθετο, είναι διαφορετικό από το κόμμα το οποίο έχει την κεντρική κυβέρνηση. Τελευταία παρατήρηση η Επιτροπή Περιφερειών ήδη από σήμερα έχει ε, κάποια εργαλεία παρακολούθησης τα οποία σας υποβάλλει έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει συγκεκριμένη απτή παρακολούθηση ε, όλων των στοιχείων. Ε, η αντίστοιχη υπηρεσία λοιπόν της Επιτροπής Περιφερειών θα σας δώσει τα στοιχεία αυτά. Όσον αφορά δε την ρήτρα επενδύσεων έχω να πω το εξής. Οτιδήποτε μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να προχωρήσει ε, πέρα από τέτοιες ε, σφιχτές διαδικασίες όπως η μακροοικονομική αιρεσιμότητα μας βρίσκει σύμφωνος. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την εργασία του και παραμένουμε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αγαστή μας συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών ε, και σας ευχαριστούμε για την συμβολή σας στη συζήτηση. Πριν δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, μάλλον αυτό θα δώσω το λόγο ε, στον κύριο Βονμπρέσκα, τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης Εκτιμάμε ιδιαίτερα το ότι η έκθεση αυτή αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις κατευθυντήριες γραμμές ακολουθεί μια πολύ συνετή προσέγγιση για την εφαρμογή του άρθρου 23. Νομίζω ότι έχει αναφερθεί αρκετά συχνά πως θέλουμε και εμείς κατά γενικό κανόνα να επιλέγουμε την σταθερότητα και όχι τις συχνούς επαναπρογραμματισμούς και να κάνουμε και μια γενική παρατήρηση. Συμβαίνει συνέχεια επαναπρογραμματισμός. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι ε, ασυνηθιστό γιατί όταν μιλάμε για περίοδους εφαρμογής δεκαετών όπου οι προτεραιότητες αλλάζουν και ότι κάποια στιγμή θέλεις και εσύ να προσαρμοστείς και να προσαρμόσεις τα προγράμματα είναι φυσιολογικό. Αυτό το οποίο προσθέτει το άρθρο 23 στις προηγούμενες διατάξεις για τον επαναπρογραμματισμό είναι πως δίνει το δικαίωμα πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή μπορεί να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ένα κράτος μέλος να επαναπρογραμματίσει μόνον όμως αν υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα οι οποίες δικαιολογούν μία περαιτέρω συγκέντρωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε συγκεκριμένη πρόκληση που να έχει εντοπιστεί σε αυτές τις συγκεκριμένες συστάσεις. Άρα λοιπόν έχουμε το βάρος απόδειξης το οποίο επιβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δικαιολογήσει οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα επαναπρογραμματισμού υποβάλλει στο κράτος μέλος. Και τότε ακόμα και στην περίπτωση αυτή η περιφέρεια και το κράτος μέλος θα επιλέξουν ε, τα μέτρα που θα χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί αυτή η σύσταση, η συγκεκριμένη σύσταση ανακράτος. Άρα λοιπόν τα μέτρα τα επιλέγουν η περιφέρεια και το κράτος μέλος μετά από ένα τέτοιο αίτημα από την Κομισιόν για επαναπρογραμματισμό. Κάνα σχόλια για συγκεκριμένα θέματα που ανέφεραν αρκετοί από εσάς σήμερα. Το πρώτο θέμα, το 6, το 8 και το 24, είναι ένα πάγιο αίτημα να προσφέρει παραπάνω πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς αυτές οι συστάσεις, η ανακράτους, θα εφαρμοστούν στα νέα, στις νέες γενναίες προγραμμάτων. Εμείς λοιπόν θα ξεκινήσουμε μια σε μελέτη φέτος, όπου θα ερευνήσουμε το πώς αυτές οι country specific recommendations, οι συστάσεις συγκεκριμένε αναχώρες στηρίζονται από τα επιχειρησιακά προγράμματα γιατί έχουμε πάνω από 300 και δεν έχουν εγκριθεί όλες χρειάζεται προσπάθεια θα ξεκινήσουμε όμως φέτος θα επανέλθουμε και θα σας τα παρουσιάσουμε Έχουμε το σημείο 11 και εμείς έχουμε τις ίδιες ανησυχίες με εσάς. Δεν θέλουμε η όλη διαδικασία να είναι υπερβολικά περίπλοκη, ε, δύσκολη και δεν θέλουμε καμία ε, επικάλυψη με τους κύκλους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Να είστε σίγουροι λοιπόν πως οι επικαλύψεις δεν θα υπάρχουν σε οποιοδήποτε έτοιμο επαναπρογραμματισμό. Τουλάχιστον δεν θα επηρεάζουν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θέλουμε λοιπόν εσωτερικές διατάξεις με προθεσμίες για τις υπηρεσίες μας, σύμφωνα με τις οποίες θα παρακολουθούμε ό,τι γίνεται σε επίπεδο αιτήματος επαναπρογραμματισμού. Για το άρθρο 14... Συμφωνούμε πως οι δημοσιονομικές πολιτικές είναι ένα θέμα που επηρεάζουν και σε εθνικό αλλά και σε χαμηλότερο επίπεδο Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς συμπεριφέρεται, ε, πώς συμπεριφέρονται όλα τα επίπεδα και πώς επηρεάζουν οι συμπεριφορές αυτές το εθνικό χρέος. Μιλάμε για κοινή ε, συμμετοχή και ενοχή όλων των ε, επιπέδων κυβέρνησης και το έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές αυτό. Πρέπει να σας πω πως δεν είναι επιλογή μας να μην αναφερόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις κατευθυντήριες γραμμές. Ο λόγος για τον οποίο δεν αναφέρθηκε είναι πως οι κατευθυντήριες γραμμές ακολούθησαν μία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2013 που αναφέρει ρητά, αναφέρεται ρητά στις πρώτες έξι παραγράφους του άρθρου 23 όπου η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι πολύ σημαντική, δεν περιγράφεται γιατί περιγράφεται στα, στις παραγράφους 15 και κάτω του άρθρου. Γι' αυτό δεν σας αναφέρουμε. Ακολουθήσαμε απλώς την σειρά που έχουμε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Δεκέμβριο του 2013. Τούτου λεχθέντος ξέρετε και εσείς πως το άστρο 23 σε πολλές ε, στιγμές αναφέρεται στην ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στον ε, δομημένο διάλογο μεταξύ των δύο, στην δίκαιη εφαρμογή του άρθρου. Άρα λοιπόν σίγουρα θα είναι πολλές οι ευκαιρίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει την άποψή του, να τη μεταφέρει για περιπτώσεις που η δράση δεν ήταν ε, αποτελεσματική ή για ενδεχόμενη αναστολή. Και βεβαίως θα σας τηρούμε ενήμερους εάν προκύξει κάποια από αυτά τα δύο. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ. Η Κομισιόν είναι σίγουρη πως οπωσδήποτε θα παρατηρούμε και θα παρακολουθούμε και θα αναμένουμε την ανάλυση σας αναχώρα και το πώς βλέπετε την συμβολή της πολιτικής συνοχής στις συστάσεις αναχώρα. Κύριε Μπλάνκο Λόπες, θέλετε να απαντήσετε. έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μου κάνατε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για το άρθρο 8 νομίζω και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν έδωσε κάποιες εξηγήσει. Πάντως στις κατευθυντήριες γραμμές για το άρθρο 23 είπατε πως λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια των κρατών μελών και του Συμβουλίου. Αυτό λέτε εσείς. Χαίρομαι πάντως που άκουσα αυτές τις εξηγήσεις. Να σας ευχαριστήσω και για τα σχόλια όλων. Η έκθεση αυτή ακολουθεί τα σχόλια όλων που συμμετείχαν στις ε, συζητήσεις μας και των σχεδόν γιατί μιλάμε για τη μακροοικονομική αρισιμότητα που προκύπτει από το άρθρο 23 ήταν κάτι το οποίο ε, για το οποίο δόθηκαν πολλές μάχες στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου και είχαμε μια ουσιαστικά ομόφωνη απόρριψη Οπότε θέλουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση να συμφωνήσουμε όσο το δυνατόν ε, περισσότεροι σε αυτά που θα προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι δύσκολο γιατί αυτή τη στιγμή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας χωρίζουν πολλά, όμως πρέπει να βρούμε έναν ισορροπημένο τρόπο. Νομίζω πως θα το πετύχουμε. Έχουμε ακόμα χρόνο για να ξεκαθαρίσουμε κάποιες απορίες και για να εμπαθύνουμε στο κείμενο και επίσης είναι και διαθέσιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλει να μας βοηθήσει και γι' αυτό την ευχαριστώ όπως επίσης ευχαριστώ τους υπολείπου συναδέλφους για τα σχόλιά τους, για τις παρατηρήσεις τους και μόλις κατατεθούν οι τροπολογίες και δούμε ποια είναι τα σημεία που έχουμε κοινά θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτή την εκκρισμό στο δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση λαμβάνοντας υπόψη επίσης και την ε, Επιτροπή Περιφερειών η οποία αναγνωρίζει πως είναι ισορροπημένη η πρότασή μας, αλλά βεβαίως έχει και αυτή τα σχόλιά της. Έχουμε χρόνο. Μπορούμε να συνεχίσουμε και να βελτιώσουμε αυτή την ε, γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου για το πώς εφαρμόζεται το άρθρο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ομάδα μας εδώ στην Επιτροπή μας που με βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε 1,5 μήνα ακόμα και με όλους όσους έχουν διάθεση να υποβάλουν τροπολογίες ή να συζητήσουμε, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την πολύ θετική συζήτηση. Να θυμίσω ότι προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών θα είναι στις 19 Μαΐου το μεσημέρι. Και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο της υπηρεσίας διατάξεων που αφορά την αρχική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή Αδριατικής και Ιωνίου. Η συγητής είναι ο κύριος Ιβάν Γιακοβτσίτς της ΑΛΔΕ μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2013 η Κομισιόν ε, δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της Ένωσης για την Αδριατική Θάλασσα και τον Ιούνιο. Τον, το Ιόνιο, συγγνώμη. Ε, πρόκειται για την τρίτη μακροπεριφερειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης για, που και αφορά χώρες στην πλειοψηφία τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και υποψήφιες χώρες όπως η Αλβανία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία. Όλοι ε, η Βοσνία Ερσεγοβίνη επίσης έχει ξεκινήσει την διαδικασία η οποία ενδεχομένως θα καταλήξει στο καθεστώς υποψήφιας χώρας. Ε, η προσπάθεια είναι να ενοποιηθεί η περιφέρεια μέσω δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης. Ε, πάντοτε ο στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι να αυξήσει την ε, ανάπτυξη αλλά και την ελκυστικότητα της περιοχής με ανάπτυξη των παρακτήων και χερσαίων περιοχών αλλά και προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων. Θα ξεκινήσουμε την αρχική συζήτηση. Έχουμε μετά, με την παρουσίαση του εισηγητού, έχουμε παρόντες και σκιώδης αλλά και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Γιάκοφτσιτς, έχετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα, θα ξεκινήσω λέγοντας ε, ότι αυτή η πρωτοβουλία η οποία προέκυψε από τη διαδικασία bottom-up όπως ήθιστε να λέμε αφορά τις τοπικές και περιφερειακές ε, αρχές ε, οι οποίες είχαν συνεδριάσει το 2010 ε, και ολοκληρώθηκαν κατά κάποιο τρόπο υπό Ιταλική Προεδρία το Νοέμβριο του προηγούμενου έτους εδώ στις Βρυξέλλες. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτής της περιοχής και της στρατηγικής που αφορά την περιοχή είναι μια στρατηγική η οποία μας ικανοποιεί έχουμε στην περιοχή αυτή και χώρες των Δυτικών Βαλκανίων οι οποίες είναι υποψήφιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αναφέρατε ήδη κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της στρατηγικής, δεν θα τα επαναλάβω. Ωστόσο θα σας πω τι έχω σημειώσει στην στρατηγική αυτή και περιμένω οι συνάδελφοι που είναι παρόντες να μας δώσουν και τις δικές τους απόψεις και παρατηρήσεις έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα τον Ιούνιο να έχουμε και την πρώτη εκδοχή αυτής της εκθέσεως. Ε, και μετά θα έχουμε την υποβολή των τροπολογιών από του συναδέλφους, τις οποίες θα μελετήσω το καλοκαίρι και ευελπιστούμε ότι τον Οκτώβριο είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη Ολομέλεια στο Στρασβούργο ότι λέω θα μπορέσουμε ε, να ε, εγκρίνουμε την έκθεση αυτή. Είχαμε λοιπόν μία πρώτη συζήτηση στο Στρασβούργο ε, πριν από λίγο καιρό μεταξύ των ε, εισηγητών. Νομίζω ότι ήταν καρποφόρα αυτή η ε, πρώτη επαφή και ο υποφαινόμενος αλλά ε, και οι σκιώδη συζητήσαμε με πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Μετά είχαμε μία σειρά διμερών συνεδριάσεων όπου οι σκιώδεις συζήτησαν μαζί μου το θέμα της έκθεσης. Νομίζω ότι το κλίμα και το πνεύμα της συνεργασίας ήταν ε, ε, καλό. Και νομίζω ότι θα καταφέρουμε τελικά να βρούμε συμφωνία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ε, ομάδων. Προσωπικά, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πρώτο μεταξύ ίσων, γιατί όλοι θα πρέπει να δώσουν τη συμβολή τους για το έγγραφο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι τρεις φορές ε, παρέστην σε συνεδριάσεις Επιτροπής Περιφερειών. Έχουν λοιπόν στην Επιτροπή Περιφερειών μία ομάδα εργασίας για τη στρατηγική της περιοχής Αδριατικής θάλασσας και Ιωνίου. Συναντήσαμε, συναντηθήκαμε λοιπόν τρεις φορές στις Βρυξέλλες και τα συζητήσαμε. Ε, εξέφρασαν την άποψή τους ε, και με τον τρόπο αυτό συμμετείχαν στην ε, επεξεργασία αυτής της εκθέσεως. Είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να συζητήσουμε και τη δική τους άποψη για την στρατηγική που θα στην περιοχή αυτή. Πρέπει να σας πω επίσης ότι εγώ έκανα επισκέψεις σε διάφορες χώρες. Συζήτησα με τον Πρωθυπουργό της ε, Κροατίας, είμαι και Κροάτης άλλωστε, ε, μίλησα με τον αντίστοιχο ε, ηγετητή του Μαυροβουνίου, τον κύριο Βούτσιτσεφ της Σερβίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπόκοβιτς ε, εκ των σκιωδών εισηγητών ε, που κανόνισε να συναντηθώ και με τον Πρωθυπουργό της Σλοβενίας. Επίσης είχα την ευκαιρία να συζητήσω τα θέματα αυτά σε ε, διαφορετικά επίπεδα στην Ιταλία και είχα και μάλιστα ε, μια συνάντηση και συζήτηση με τον ε, επικεφαλής της περιφέρειας Βενέτσια Τζούλια. Όσον αφορά την ε, Ελλάδα θα συναντηθώ και εκεί με διάφορους υπουργούς όσον ούπο και θα μου δώσουν τη δική τους άποψη θα υπάρξει μια διάσκεψη στην Ελλάδα σχετικά με την στρατηγική της Αδριατικής θάλασσας και Ιωνίου. Όμως θα γίνει ταυτόχρονα, συμπίπτει δηλαδή, με την Ολομέλα του Στρασβούργου και θα, δεν θα έχω τη δυνατότητα προσωπικά να παραστώ, αλλά θα στείλω αντιπρόσωπο. Τι μπορώ να σας πω όσον αφορά τη στρατηγική για την περιοχή Αδριατικής Ιωνίου. Μπορώ να σας πω ότι όλοι περιμένουμε πολλά από αυτή τη στρατηγική. Ευελπιστώ πραγματικά ότι ε, θα ολοκληρωθεί με επιτυχία η στρατηγική αυτή και ότι θα δώσει τη δυνατότητα να λυθούν συγκεκριμένα προβλήματα ε, που μπορεί να αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα και που μπορεί να φτάσουν ε, σε θέματα όπως η ενέργεια, τα ε, θέματα που συνδέονται με τη θάλασσα, με την αλληλεία, με τις μεταφορές και ένα σωρό άλλα. Ευελπιστώ πραγματικά ότι θα γίνει αποδεκτή η έκθεση και στις εμπλεκόμενες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε ε, Γιάκοφτσίτς ε, για την προετοιμασία που έχετε κάνει μέχρι τώρα όσον αφορά την εκπόνηση της εκθέσεως. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τους σκιώδεις. Κύριε Μπόγκοβιτς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Τσίτσι για την εισαγωγή που έκανε, μας είπε το τι έχει γίνει σε αυτόν τον τομέα για την στρατηγική Αδριατικής ε, Ιωνίου μεγάλη περιοχή με 70 εκατομμύρια ανθρώπους συμπεριλαμβάνει την Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία και Ελλάδα ε, από τα κράτη-μέλη αλλά και κάποιες ε, χώρες ε, της ε, Ιουγκοσλαβίας, τη Σερβία Μαυρομούνια δηλαδή, τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και τα λοιπά. Μεγάλη περιοχή λοιπόν. και βεβαίως κάποιες περιοχές είναι αρκετά ανεπτυγμένες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και κάποιες άλλες είναι κάτω από αυτόν κατά 30% κάτω και το ποσοστό ανεργίας επίσης ποικίλει από 4 μέχρι και 30% υπάρχουν πολλά νησιά με άσχημες ε, διασυνδέσεις ε, και άρα υπάρχουν και προβλήματα. Η στρατηγική αυτή ξεκινάει ταυτόχρονα με την επόμενη προγραμματική περίοδο της πολιτικής συνοχής και θα πρέπει να την συμπληρώσει Η συνεργασία δεν ήταν πάρα πολύ καλή, υπήρχε και πόλεμος και όπως ήδη είπα υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαφορές αλλά και άλλες προκλήσεις Υπάρχουν κάποια λιμάνια, το Κόπερ, η Ριέκα, λιμάνια τα οποία μπορούν να μειώσουν τις διαδρομές σε σχέση με τα λιμάνια της ε, Βόρειας Ευρώπης που είναι 3.000 χιλιόμετρα βορειότερα. Αλλά βεβαίως οι οδικές ε, συνδέσεις με την ενδοχώρα είναι προβληματικές και χρειάζονται. Άρα επενδύσεις. Και βεβαίως ε, και ο τομέας ε, της ε, ενέργειας είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει για καλύτερες διασυνδέσεις. Εδώ πέρα μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παροχή φυσικού αερίου είναι κάπως προβληματική. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα που σχετίζονται με την ε, ενέργεια και με την ε, έρευνα για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο και κάποιοι θεωρούν πως υπάρχει ένας μεγάλος ε, κίνδυνος. Υπάρχουν προβλήματα λοιπόν γιατί η Αδριατική είναι κάπως κλειστή θάλασσα. Υπάρχουν προβλήματα με τα απόβλητα που δεν έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία αλλά και άλλα νερά που φεύγουν μαζί με τα νερά της ε, Σεντίνας αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τις δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, Γι' αυτό χρειάζεται νομίζω και κάποια διεθνής ε, βοήθεια. Θα πρέπει λοιπόν να απαντηθούν κάποια θεσμικά ζητήματα. Η διαφθορά είναι ένα μεγάλο θέμα. Η συνεργασία πρέπει να βελτιωθεί και να καταπολεμήσουμε και την διεθνή κλιματικότητα λοιπόν συνολική στρατηγική και άρα χρειάζεται καλύτερη συνεργασία, συντονισμός, Κάτω που έχει μεγάλη σημασία και για τα κράτη εκείνα που δεν είναι ακόμα κράτη-μέλη. Θεωρώ πως όπως είπε ο κύριος ε, Γιακοβτσίτς ε, πρέπει να προωθεί αυτή η στρατηγική. Ελπίζω να εγκριθεί λοιπόν το φθινόπωρο. Έχουμε καταθέσει και κάποιες ε, τροπολογίες για να υλοποιηθούν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γιουφρίντα, θέλετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω ότι συμμερίζομαι πλήρως τα όσα είπε ο συνάδελφος Γιάκοφτσιτς. Ε, και μάλιστα χαιρετίζω την τροπή που έχει εξ αρχής ε, πάρει η εργασία του. Είναι μια ε, έκθεση η οποία ξεκίνησε από κάτω προς τα πάνω και έτσι πρέπει να συνεχίσει. Πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρή η εργασία που από κοινού ξεκινούμε γιατί η έννοια της στρατηγικής είναι ακριβώς η υπέρβαση των εθνικών συνόρων. Είναι ακριβώς να δούμε τα εδάφια αυτά ε, βάσει των χαρακτηριστικών τους, των δομικών τους ε, χαρακτηριστικών. Έχουμε μια στρατηγική που έχει κοινό παρονομαστή δύο πελάγοι, ε, την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος. Πρόκειται για δύο θάλασσες οι οποίες είναι ιδιαίτερες και εξαιρετικά πλούσιες, αλλά που μπορούν ταυτοχρόνως να αποτελέσουν πρόσκομα και όσον αφορά την κινητικότητα και όσον αφορά την ανάπτυξη. Η στρατηγική, το είπε και ο προλήσας συνάδελφος, αφορά περισσότερο από 70 εκατομμύρια ε, ανθρώπους. Μιλούσαμε προηγουμένως για τις τρεις βασικές στρατηγικές ε, με τις οποίες το Κοινοβούλιο και η δική μας ε, Επιτροπή τις οποίες συζητάει το Κοινοβούλιο και τις και η Επιτροπή μας και πραγματικά εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Πρόκειται για μια στρατηγική η οποία εμπλέκει 8 χώρες και μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικά καλές σχέσεις ανάμεσα σε χώρες οι οποίες ήδη ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες που δεν ανήκουν ακόμα. Ε, θα πρέπει να βασιστούμε στα θετικά στοιχεία, θα πρέπει να μοιραστούμε ε, τις, ε, ε, το, τον πλούτο αλλά και να δοθεί η δυνατότητα να ε, ε, υπερβούν ε, όπου υπάρχουν και σε όποιες χώρες αυτό διαπιστώνεται, να υπερβούν λέω οι χώρες αυτές τις αδυναμίες διακυβέρνησης. Επομένως είναι σωστός ο δρόμος που ξεκινούμε και θα πρέπει η στρατηγική να ενοποιήσει κατά κάποιο τρόπο θάλασσες, παράκτιες περιοχές, εσωτερικές πλωτές οδούς. Πρόκειται για πολιτικές οι οποίες έχουν ξεκινήσει τμηματικά μέχρι τώρα και οι οποίες δεν έχουν καταφέρει τουλάχιστον να ε, βοηθήσουν στην υπέρβαση των ε, αδυνάμων σημείων των περιοχών αυτών. Εδώ τώρα πρέπει να έχουμε δύο στόχους. Πρώτος στόχος κατά την άποψή μου ε, θα πρέπει να είναι να υπάρξουν διορθωτικά ειδικά ε, μέτρα να εξυγιανθούν ε, αυτά τα, ε, έχουν, αυτά τα μέτρα τα οποία ενδεχομένως έχουν ληφθεί και τα οποία έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Ας πούμε να λυθούν προβλήματα κατάχρησης της δόμησης όπως ας πούμε και οτιδήποτε άλλο αρνητικό πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα ας πούμε επίσης όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αλληλείς και που ε, κάποιες αρχές ε, ε, περιοριστικές που διέπουν την αλληλεία τις αισθάνονται ως ιδιαίτερα περιοριστικές για τους, για τους ίδιους. Επίσης θα πρέπει να δοθεί μια νέα όθηση μέσω των μεγάλων έργων, μέσω της διασύνδεσης αλλά και μέσω, των, μέσω της έρευνας. Ξέρουμε ότι υπάρχει η μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιωνίου ε, που θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, αναπτυχθεί μέσα από τους ε, τρεις πυλώνες που έχουμε ήδη καθορίσει για την περιφέρεια αυτή. Και εδώ αναφέρομαι στην ανάπτυξη και κυρίως στην όθηση που μπορούν να έχουν και το ρόλο το μεγάλο μπορούν να παίξουν ακαδημίες, πανεπιστήμια, κέντρα έρευνας. Καταλαβαίνετε ότι γύρω από αυτούς τους πυλώνες ε, θα πρέπει να περιστρέφεται ο δικός μας άρτος επίουσιος, η δικιά μας καθημερινή δουλειά που είναι η πιο πολιτική δουλειά. Ε, υπάρχει όμως και ένας τέταρτος πυλώνας ε, η ποιότητα του περιβάλλοντος, ε, κάποιες παρεμβάσεις ε, που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να κάνουμε όσον αφορά περιοχές ε, οι οποίες θα πρέπει να αναπτύξουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές ε, ε, περιοχές ε, όπου θα πρέπει να κινητροδοθεί οπωσδήποτε υπεραιτέρω έρευνα έτσι ώστε να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις και έτσι ώστε να υπάρξει και η σωστή πρόληψη. Ε, φυσικά θα πρέπει να αναφέρουμε και την έρευνα όσον αφορά ε, την χρήση πράσινης ενέργειας, νέων μορφών ενέργειας. Και βεβαίως υπάρχει το μεγάλο κεφάλαιο των μεταφορών, διασύνδεση των περιοχών, γιατί εδώ έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχουμε προβλήματα όσον αφορά την εδαφικότητα της περιοχής, όσον αφορά τις υποδομές της περιοχής και να μην λησμονούμε βέβαια και το κεφάλαιο ε, το οποίο αφορά αυτό το δίκτυο ε, το οποίο θα πρέπει να συνδέσει τους λιμένες και τους αερολιμένες έτσι ώστε η κινητικότητα ε, να γίνει ολοκληρωμένη και αποτελεσματική. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ ε, μιλώντας ακόμα περισσότερο για να αναφερθώ στον τουρισμό και τον αηφόρο τουρισμό. Ξέρουμε ότι η περιφέρεια έχει αριθμεί ορισμένα από τα τμήματα της ε, Ευρώπης ε, και επομένως ε, θα πρέπει οπωσδήποτε στα πλαίσια της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις περιοχές αυτής της περιφέρειας είναι πραγματικά περιοχές οι οποίες καλύπτονται από την UNESCO θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση τους. Φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν ε, με προσεκτική χρηματοδότηση, με ικανή και αρκετή χρηματοδότηση. Η στρατηγική θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, θα πρέπει να είναι καλά χρηματοδοτημένη ε, και οπωσδήποτε θα πρέπει να πατάει σε μια καλά διαρθρωμένη ε, λογική στρατηγική. Εν συμπεράσματι, κατά την άποψή μου, η εργασία που μας περιμένει είναι μεγάλη, είμαστε όλοι διατεθειμένοι να δουλέψουμε, είμαστε όλοι διατεθειμένοι ε, να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε σε αυτό που θα πρέπει να είναι μια συνολική προσέγγιση ε, και που θα πρέπει να απορρέει αυτή η προσέγγιση από ε, μακρόπνοα σχέδια, γιατί θέλουμε να ενεργήσουμε με τρόπο ώστε τα μειονεκτήματα να μετατραπούν σε πλέον εκτήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ φιλόδοξη η πληροφοριών. Λοιπόν, κύριε Τόμασιτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση και τιμή το ότι είμαι σκιώδη Υγήτρια και βοηθά του συναδέλφου στην σύνταξη αυτή της στρατηγική. Θεωρώ πως ε, θα μπορούσε να έχει έναν πάρα πολύ καλό αντίκτυπο στις χώρες της ε, Αδριατικής ε, και του Ιωνίου. Έχουμε λοιπόν τέσσερις πυλώνες οι οποίοι πρέπει να ισχύσουν παράλληλα. Επίση, πρέπει να τονίσουμε πω το σχέδιο δράση τη ε, Κομισιόν δεν είναι δεσμευτικό, ούτε και η στρατηγική. Πρόκειται απλά για μια πρόταση για το πώ θα ε, έχουμε κάποια πρόοδο και θα συνδεθεί αυτή η περιφέρεια. Επίσης ε, γίνονται κάποιες προτάσεις για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους υφιστάμενους πόρους. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ενημερώσουμε το κενό και τους ενδιαφερόμενους για τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτή η στρατηγική σωστή ε, εφαρμογή της στρατηγικής εξαρτάται από τις ε, χώρες και την δυνατότητα που έχουν να απορροφήσουν τα κονδύλια. Θα πρέπει λοιπόν να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό για να έχουμε επαρκή απορρόφηση των κονδυλίων και διοικητική ικανότητα. Ο δεύτερος πυλώνας, η διασύνδεση της περιφερειας είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί περιέχει διάφορες επιλογές για ανάπτυξη. Είναι άσχημα διασυνδεδεμένη περιοχή της Αδριατικής ε, σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Παραδείγματο χάρη, εάν ναι, θέλω να πάω σε ένα νησί από το Ζάγκρεμπ χρειάζομαι 9 ώρες. Μιλάω εδώ πέρα για το δικό μου το νησί βεβαίως, οπότε πιο γρήγορα πάω στον Καναδά, το Κότοκο πιο γρήγορα πάω στον Καναδά παρά στο νησί μου. Λοιπόν, οι μεταφορές ε, και τα ενεργειακά δίκτυα είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την κοινωνική ανάπτυξη. Επίσης είμαι και κατά της εξόριξης πετρελαίου στην Αδριατική. Πρόκειται για απειλή για τον τουρισμό που είναι πολύ σημαντικό τομέα της κροατικής οικονομίας. Επίσης κινδυνεύει και η αλληλεία που επίσης παρέχει θέσεις εργασία ολόκληρο το χρόνο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις περιοχές εκείνες όπου δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες απασχόλησης, π.χ. νησιά και μικρές παραθαλάσσιες πόλεις. Δεν βλέπω τον κύριο Παπαδημούλη. Λοιπόν, κύρια Βάρνερ, έχει τον λόγο. Thank you, Madam Chair. I have to apologize. Our Green Shadow. Uh... Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, κύριος ε, Ντάβορ ε, έχει κάποια άλλη υποχρέωση. Να αναφέρω αυτά τα οποία απασχολούν τους πράσινους. Αναφέρθηκαν ήδη η εξόρυξη πετρελαίου στην Αδριατική. Ξέρετε πως ε, η κυβέρνηση της Κροατίας έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για εξόρυξη πετρελαίου και ενέκρινε διάφορα πεδία υπεράκτια πεδία έρευνας με τρόπο πάρα πολύ γρήγορο και μη διαφανή Τίθεται λοιπόν ζητήματα συμμόρφωση με την νομοθεσία, έλλειψη δημόσια συζήτηση και βεβαίω ω πράσινοι εμεί πρέπει να πούμε πως ε, κινδυνεύει όχι μόνο η θαλάσσια βιοπικιλότητα και το εξαιρετικό οικοσύστημα, αλλά όπως υπόθηκε ήδη και η δουλειά εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν από τον τουρισμό και την αλληλεία. Οπότε θα θέλαμε να έχουμε κάποιες ε, έντονες διατυπώσεις κατά αυτών των αποφάσεων και ελπίζουμε η συγκήτρια να μας εισακούσει γιατί όπως είπαμε θα πρέπει να βασιστούμε στους τέσσερις πυλώνες γαλάζια ανάπτυξη, αηφόρος τουρισμός, διασύνδεση των περιφερειών και βεβαίως ποιότητα του περιβάλλοντος. Και εδώ πέρα το πετρέλαιο, τα απειλή και τα τέσσερα αυτά. Σας ευχαριστώ κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για το προσχέδιο. Θα ξεκινήσω εκφράζοντας την ικανοποίησή μου για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ε, η οποία αφορά μια μακροπεριφέρεια 70 εκατομμυρίων κατοίκων, συνδυάζει ε, ε, χώρες μέλη και χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένω βέβαια και το πραγματικό προσχέδιο έτσι ώστε να δώσω μια πιο συγκεκριμένη γνωμοδότηση, αλλά προς στιγμή μπορώ να πω ότι αυτοί οι τέσσερις πιολώνες που έχει επιλέξει είναι σωστοί. Ε, ε, αλλά βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες ε, των χωρών γιατί δεν έχει έννοια ε, να αναφερθούμε ας πούμε στην ε, ανάπτυξη ενός συστήματος μεταφοράς ενέργειας που όμως δεν θα λαμβάνει υπόψη ας πούμε τα οικοσυστήματα γιατί υπάρχουν ήδη συστήματα όπως τα τεμπαρόσα και άλλα τάπ και λοιπά τα οποία αφορούν το Ιόνιο. Είναι άλλες έξι επιτροπές οι οποίες θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό αυτό και ακριβώς ευελπιστώ ότι μέσα στα πλαίσια μιας εγκάρσιας αντιμετώπισης θα μπορέσουμε να δουλέψουμε. Ε, είναι πολλές, ε, πολλά τα διακυβεύματα για την περιφέρεια. Ε, αναφέρομαι εδώ εν είδη παραδείγματος στην ανάπτυξη ενός οικοβιώσιμου μοντέλου ας πούμε το οποίο μας είναι ιδιαίτερος προσφυλές και εμείς ε, θα αποφασίσουμε ε, ποια θα είναι η πορεία, η κατεύθυνση που θα δώσουμε σε αυτήν την πολύ σημαντική έκθεση μέσω των τροπολογιών που θα υποβάλουμε στον συνάδελφο στα πλαίσια μιας ε, συνεργασίας που εύχομαι να είναι παραγωγική και καλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σουίκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα το πω ανοιχτά. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, είμαι εδώ στη συνεδριάση, είμαι μέλος της ΑΦΕΤ και της Επιτροπής ΕΜΒ. Και επειδή ακριβώς χρειάζεται να συντάξω τη γνωμοδότηση, ήθελα να ακούσω τι θα πείτε κι εσείς στη δική σας Επιτροπή για το θέμα γιατί μόνο τότε θα είμαι σε θέση να ρωτήσω Ο κύριος Γιάκοψης και εγώ συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια όταν στήθηκε αυτή η μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου, ε, ήλπιζα πως το έγγραφο σήμερα θα συμπεριλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες αλλά ξέρω πως ε, πολλά ακόμα βρίσκονται στα σκαριά. Ίσως θα έχω περισσότερες ε, ε, πληροφορίες να δώσω αφού συζητήσω και με τη συνάδελφο από την Ιταλία. Πάντως υπάρχει ένα εγγραφό το οποίο προετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει τη μορφή της ανακοίνωσης, απευθύνεται στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών και έχουμε τρία κράτη τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της ε, Αδριατικής Ιωνίου και που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σημείο ε, είναι αυτό στο οποίο πρέπει περισσότερο να σταθούμε λόγω των εξελίξεων που είναι η μετανάστευση στη Μεσόγειο να σας πω πως πολύ σύντομα όλα αυτά θα περάσουν και θα επηρεάσουν και την λεκάνη της ε, Αδριατικής και του Ιωνίου άρα λοιπόν θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε τα θέματα αυτά και στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Κάποιοι είπαν πως στο παρελθόν αποτελούσαν εμπόδιο οι θάλασσες. Όμως για το Ιούνιο και την Αδριατική πρέπει να σας πω πως η θάλασσα πάντα αποτελούσε μια γέφυρα. Ίσως σήμερα ενδεχομένως να αποτελούν πρόβλημα. Όμως εγώ επειδή είμαι από το νότο της Κροατίας, είμαι από τον Ντουμπρόβνικ, πρέπει να σας πω πως για να πάω από τον Ντουμπρόβνικ στη Ραβένα πόλη με την οποία έχουμε αδελφοποιηθεί. Πρέπει να πάω πρώτα στο Ζάγκρεπ, μετά να πάω στη Λιουμπιάννα από εκεί να πάω στην Πολόνια και από εκεί να κατέβω στη Ραβένα, ενώ είναι ακριβώς απέναντί μου ε, αν απλώς διασχίσω την Αδριατική. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε στο μέλλον, να επιτρέψουμε μια νέα ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας με τον τρόπο αυτό. Μια στρατηγική λοιπόν μας χρειάζεται, η οποία όμως θα εφαρμοστεί, γιατί υπάρχει στρατηγική σε επίπεδο εγγράφου, το έστειλε σε εμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει όμως να δώσουμε σάρκα και οστά, να αναθέσουμε καθήκοντα στα κράτη-μέλη, γιατί διαφορετικά η στρατηγική αυτή δεν θα εφαρμοστεί. Όπως σας είπα, είμαι από την Κροατία. Αυτές οι κροατικές ακτέ. Για το θέμα λοιπόν της εξόρυξης πετρελαίου δεν είμαστε απριόρι υπέρ ή κατά. Αυτό το οποίο δεν μας ικανοποιεί είναι αυτό το οποίο κάνει η κρατική κυβέρνηση σήμερα που ε, έχει επιτρέψει εξορίξεις χωρίς καμία μελέτη και χωρίς να δημοσιοποιεί ε, τα στοιχεία που έχει ε, στο ευρύ κοινό. Εμείς θέλουμε διαφάνεια. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους και με τους πράσινους και με την κυρία Τόμασιτς που θεωρούν πως αυτό είναι από τα πιο σημαντικά θέματα στα βόρεια ύδατα της Αδριατικής. Επαναλαμβάνω, χαιρετίζω το γεγονός πως γίνεται αυτή η συζήτηση. Έχουμε κάποιες προθεσμίες στις διάφορες επιτροπές μας για τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων. Νομίζω όμως πως πριν προχωρήσουμε στη σύνταξη γνωμοδότηση χρειαζόμαστε ένα σχέδιο στρατηγικής και κατόπιν μια γνωμοδότηση πάνω στο σχέδιο αυτό. Καλύτερο συντονισμός λοιπόν μεταξύ των επιτροπών μας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την δουλειά μας, αντιλαμβανόμαστε πόσες συνεδριάσεις έχουν ήδη οργανωθεί. Κύριε Βαλκαρσέλ, θέλετε να μιλήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από τρία χρόνια ο κύριος Αλφονσίν ξεκίνησε τη συζήτηση για το αν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μία μακροπεριφέρεια στη Δυτική Μεσόγειο. Και αυτό χωρίς να ε, έρθουμε σε ανταγωνιστική σχέση με την Ένωση για τη Μεσόγειο. Και όταν τελείωσε ε, τις προσπάθειες αυτές, παρόλο που ακούστηκαν κάποιες επιφυλάξεις, πολλές περιφέρειες είπαν πως ναι, μας ενδιαφέρει το θέμα και θέλουμε να συνεχίσουμε. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν να συνεχίσουμε να κάνουμε περισσότερες μελέτες και και διαθεσμική συνεργασία όπως ακριβώς προτείνεται μέσω αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας πρωτοβουλίας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πως τα ε, φρικτά γεγονότα σε, στην ε, περιοχή αυτή εντείνουν τα αισθήματά μας πως το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στη Μεσόγειο και πως τα προγράμματα συνεργασίας αυτή τη στιγμή είναι άσχημα διαστρωμένα και πολύ δύσκολα επιτρέπουν το να λειτουργήσουμε σωστά και να κάνουμε ε, τα κατάλληλα βήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα ήταν ε, μάλλον αρνητική για την ε, ανάπτυξη αυτών των μακροπεριφερειών και αυτών των ε, πρωτοβουλών. Είδαμε όμως πως αποτελεί μια προστιθέμενη αξία για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική συνοχή και ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν αυτές οι δυνατότητες να ανοίξουν και για άλλες περιφέρειες. Κάθε στρατηγική κυρία Πρόεδρε που μπορεί να συνεισφέρει στο να δημιουργήσει μεγαλύτερη περισσότερη συνεργασία μεταξύ περιφερειών και που θα ενθαρρύνει έργα που θα ενδυναμώσουν τις οικονομίες των χωρών μας είναι καλοδεχούμενες. Εφόσον βέβαια δεν θα δημιουργήσουμε ε, παραπάνω γραφειοκρατία από ό,τι έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις... Α, ο κύριος Βανλής Ρόι. <clears throat> Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω μια εξαιρετική συζήτηση και θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το επιπρόσθετο που προσφέρουμε με αυτή την έκθεση. Έχει διάφορα θετικά κεφάλαια και πρέπει να δούμε την διακυβέρνηση και την συνεργασία που υπάρχει γιατί μπορεί ο καθένας να κάνει το δικό του αλλά αν τα συγκρίνει με τους άλλους θα πει ότι δεν έχω καταφέρει πολλά οπότε ποιο είναι το αποτέλεσμα που κάνατε ε, της εξέτασης ε, αυτής Και βεβαίως ε, αυτό είναι το οποίο θα οδηγήσει σε καλύτερο αποτέλεσμα. Δεύτερον, για το θέμα αυτό της διοίκησης. Υπάρχουν πάρα πολλά δημιουργικά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν διασυνοριακά. Το είδαμε αυτό και στην Βαλτική παραδείγματος χάρη που ήταν η πρώτη περιφέρεια στην οποία υπήρχε αυτή η συνεργασία. Αλλά εκεί πέρα χαρακτηρίζαν κάποιες προτεραιότητες. Δεν ξεκινήσαμε με όλα τα πράγματα μαζί. Είπανε οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα να καθαρίσουμε λίγο την θάλασσα. Τη στιγμή λοιπόν που ξεκινάς να κάνεις κάτι τέτοιο έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και μετά κοιτάς Είσαι διατεθειμένος να λάβεις τα μέτρα που χρειάζονται για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Έτσι γίνεται. Δηλαδή πρέπει να φτάνουμε στον πυρήνα του προβλήματος και όχι μόνο να μιλάμε, αλλά να πούμε πως πρέπει να, γίνει, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα διαφορετικά. Και έτσι θα έχουμε πραγματικά μία προσθέμενη αξία της στρατηγικής αυτής. Αυτό θέλω να ακούσω. Πού υπάρχει. Και τέλος, αυτό το οποίο λέω συνέχεια, ο ίδιος δίσκος που παίζει συνέχεια. Δεν υπάρχει επιπρόσθετη χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχή στις μακροπεριφέρειες. Αν κάνουμε κάτι τέτοιο διαλύουμε την περιφερειακή μας πολιτική. Πάρα πολύ απλά. Αν η Ευρώπη επιλέξει τις μακροπεριφέρειες. Ε, ας κάνουμε, τα, ας πάρουν τα κράτη-μέλη την θέση των περιφερειών. Δεν θα γίνει λοιπόν κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε λίγο βαθύτερα στο ποια αποτελέσματα μπορείτε να έχετε. Αυτό θα ήθελα λοιπόν εγώ να δω, ένα τέτοιο έγγραφο που θα περιγράφει την προστιθέμενη αξία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γιάκοβτσίτς, έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να ακούσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον κύριο Μπαλέτε. Έχετε τον λόγο. Ναι, Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος επιτρέψατε μου να πω πως αναμένουμε την έκθεση η οποία συντάσσεται και η συζήτηση νομίζω έδειξε πως θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο είπαν αρκετοί βουλευτές. Η στρατηγική αυτή είναι, μια προσέ... είναι αποτέλεσμα προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω. Το σχέδιο δράσης που είναι κομμάτι της ε, στρατηγικής ε, Αδριατικής Ιουνίου είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης διαβούλευσης με τοπικές εθνικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών, και όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους μπορέσαμε να βρούμε σε 10 μήνες το 2013, αρχές του 2014. Το περιεχόμενο λοιπόν τέσσερις πυλώνες είναι αποτέλεσμα της διαβούλευσης που με βάση τα μαθήματα που αντλήσαμε από τη Βαλτική και τον Δούναβη είναι πολύ εστιασμένοι. Εστιασμένοι σε τέσσερις πυλώνες που αναγνώρισαν οι ενδιαφερόμενοι ως τους πιο σημαντικούς και ήταν η συνεργασία μεταξύ χωρών και περιφερειών που θα έδιναν την μεγαλύτερη προστέμενη αξία. Δηλαδή η μπλε οικονομία, διασύνδεση περιφέρειες, ε, περιφερειών και ενεργειακών δικτύων ποιότητα του περιβάλλοντος και βιώσιμος τουρισμός. Οι δράσεις λοιπόν είναι ενδεικτικές θα έλεγα όπως υπόθηκε και παραδείγματα κοινών έργων. Αλλά οι τέσσερις πυλώνες, οι οχτώ χώρες συμφώνησαν να ξεκινήσουν τους τέσσερις πυλώνες μόνο. Οπότε νομίζω πως ε, είναι πολύ εστιασμένοι πρωτοβουλία και ελπίζουμε η έκθεση να βοηθήσει ακριβώς ε, στην εστίαση αυτή για να μπορεί να έχει αποτελέσματα η στρατηγική αυτή. Το δεύτερο που θα ήθελα να αναφέρω είναι πως είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για αυτή την στρατηγική. Είμαστε στη βάση στην οποία περνάμε από τα λόγια στις πράξεις. Η στρατηγική υιοθετήθηκε το φινόβορο μας πέρασε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είχαμε μια αρχή εκδήλωση στις 18 Νοεμβρίου ε, επί Ιταλικής Προεδρίας και έκτοτε συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με εθνικές ε, και περιφερειακές αρχές για να δημιουργήσουμε κάποιες δομές διοίκησης. Αυτή ήταν η καμπή την οποία ανέφερα. Δεν ήταν εύκολο, δεν γίνεται αμέσως, απαιτείται μια προσπάθεια από όλους τους ενδιαφερόμενους ακριβώς για να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Για να δημιουργήσουμε αυτές τις δομές οι οποίες πράγματι θα φέρουν αποτελέσματα. Οι οχτώ χώρες ε, θα έλεγα είναι οι διοκτήτες αυτής της στρατηγικής, η διοίκηση θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη σε επίπεδο τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών. Η Κομισιόν θα βάλει κάθε προσπάθεια για να συνεχίσει να συντονίζει τη στρατηγική αυτή αλλά όπως σας είπα την στρατηγική την ασκούν οι 8 χώρες. Όπως είπα λοιπόν αναμένουμε την έκθεση που θα υιοθετηθεί από την Επιτροπή σας τον Ιούνιο. Είμαστε έτοιμοι για να συνεισφέρουμε, να βοηθήσουμε εάν ζητηθεί η βοήθειά μας και ελπίζουμε η έκθεση αυτή να βοηθήσει ακριβώς ε, στην καμπή στην οποία βρισκόμαστε στο να κινητοποιηθεί η εθνική και η περιφερειακή διοίκηση στην φάση της εφαρμογής για να αρχίσει να έχει αποτελέσματα η στρατηγική αυτή. Καθώς υπάρχουν πολλές προσδοκίες και δικαίως στην περιοχή. Ευχαριστώ θα έχουμε ενδεχομένω την ε, έκθεση τον Ιούνιο, θα τη συζητήσουμε σε μια συνεδρίαση ε, της Επιτροπής μας και ενδεχομένως η συζήτηση για τις ε, ε τροπολογίες ε, θα γίνει τον Ιούλιο. Κύριε Γιάκοφ, σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον κύριο Βαν Χίστερόι για τις ερωτήσεις του. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να εξηγήσω μερικά έτσι, γενικά στοιχεία. Ε, οι στρατηγικές ε, για τις μακροπεριφέρειες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης έχουν ένα σημείο έναρξης είναι, ε, είναι στην ουσία τρεις αρνήσεις, ε, δηλαδή ε, άρνηση για επαναπρογραμματισμό, άρνηση για νέες χρηματοδοτήσεις, άρνηση για επιπλέον δομές. Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς οι κανόνες είναι αυτοί που είναι και επομένως και για την περίπτωση Αδριατικής Ιωνίου δεν θα αλλάξουν. Ε, επίσης εγώ κατανοώ απολύτως αυτά που λέτε αλλά δυστυχώς ε, δεν μπορώ να εφεύρω οτιδήποτε. Υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχουν κανόνες και πρέπει να τους ε, σεβαστούμε. Βεβαίως μπορούμε να προσπαθήσουμε να τις αλλάξουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε την πολιτική αυτή των τριών αρνήσεων ε, με, και να την αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο και τότε οπωσδήποτε θα τροποποιηθεί αναλόγως και η στάση μας. Ας επανέλθουμε στο θέμα μας. 70 εκατομμύρια άνθρωποι από 8 χώρες. Αυτή η στρατηγική είναι πάρα πολύ σημαντική για την Νότια Ευρώπη. Ιδίω δε στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποια νέα ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά με τον κύριο Παπαδημούλη ήδη έχουμε συζητήσει το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί το θέμα των μετα... της μετανάστευσης. Ε, η μετανάστευση και τα συνεπακόλουθα προβλήματα για την Ιταλία, ε, συγγνώμη για την Ελλάδα αλλά και για άλλες συμμετέχουσες χώρες είναι κάτι το οποίο και κατά τη δική μου άποψη θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ε, έκθεση. Άσχετα από το γεγονός ότι ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τέσσερις ε, πυλώνες ε, στους οποίους δεν έχει περιληφθεί το θέμα της μετανάστευσης. Κάτι άλλο τώρα. Η στρατηγική αυτή έχει τεράστια προστιθέμενη αξία διότι στην ουσία δίνει την δυνατότητα ε, να διασυνδεθούν οι ε, συμμετέχουσες ε, χώρες. Η κυρία έτσι το είπε, πιο εύκολα φτάνει από εδώ στον Καναδά παρότι στο δικό της το χωριό θυμάμαι ότι μια φορά ήθελα να πάω στην Πεσκάρα και έπρεπε να κάνω κάτι ακροβατικά, να πάω από το Ζάγκρο στη Ρώμη και από τη Ρώμη στην Πεσκάρα και καταλαβαίνετε ε, η απόσταση ε, και Ζάγκρεβ-Πεσκάρα είναι κάτι ως 100 μίλια. Επομένως υπάρχει σαφές πρόβλημα διασύνδεσης της περιοχής. Αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε εδώ είναι ε, μία ισχυρότερη διασύνδεση της ε, περιφέρειας. Αυτό δεν ε, αφορά μόνο τα κράτη-μέλη της Ένωσης, αλλά όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην ε, περιοχή. θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Ε, υπάρχουν ε, ήδη χώρες οι οποίες ε, είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένες. Επίσης πριν από την περιοχή Αδριατικής θάλασσας και Ιωνίου υπήρχε ήδη μία οργάνωση η οποία συνέβαινε την περιοχή και που ήταν πολύ δραστήρια. Αλλά τώρα θέλουμε να έχουμε πραγματική προστιθέμενη αξία και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε. Και επομένως εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καλό πλαίσιο για την μελλοντική συνεργασία όχι μόνο μέσω και βάση της ε, πολιτικής συνοχής αλλά και άλλων εργαλείων. Ο ε, πρόεδρος Γιούνκερ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν και να στηρίξουν αυτήν την στρατηγική. Ε, κύριε Βανίστερο, θα σας ζητήσω να με προσέξετε λίγο γιατί θα απαντήσω τώρα στην ερώτησή σας. Συγγνώμη που σας διακόπτω από αυτό που κάνατε. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό ε, ότι ο κύριος Κατάινεν είναι διατεθειμένος, είναι πρόθυμος να είναι ειλικρινής. Τον ρώτησα άμεσα ε, εάν τα, ε, τα χρήματα ας πούμε του Ταμείου Γιούνκερ ε, θα πάνε και προς την περιοχή Αδριατικής Ιωνίου και προς χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου απήντησε ναι, εάν υπάρχει αποδεδειγμένο συμφέρον εταιριών από χώρες μέλη στην περιοχή αυτή, ας πούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από σλοβενικές, σουηδικές ή άλλες εταιρείες. Ε, επομένως ε, είναι σημαντικό να... Ε, υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Είναι το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ενέργεια των υδάτων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην περιφέρεια αυτή κυρίως μέσα στα πλαίσια της ε, οικονομίας ε, με χαμηλή χρήση, ε, χαμηλή χρήση άνθρακα και χαμηλό διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής. Επίσης η παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι σημαντική. Με ρωτήσατε στο Στρασβούργο εάν προτίθεται να συμμετέχει χρηματοδοτικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τα ε, ε, προγράμματα ε, διασύνδεσης των διαφόρων περιοχών της Αδριατικής Ιωνίου. Ας πούμε αναφέρομαι στον διάδρομο της Αδριατικής ή το, ο, ο αγωγός αερίου που θα πρέπει να ακολουθήσει ενδεχομένως έναν από τους διαδρόμους ή ενδεχομένως ο εξυγχρονισμός του ε, ε, σιδηροδρόμου και η νέα ε, χάραξη σταθερά στροχιάσα Αγκώνα Μπάρι. Όπως ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που προέρχονται από τις συμμετέχουσες χώρες. Εν συμπεράσματι θα ήθελα να πω τα εξής. Δεν θέλω να μακρηγορώ, αλλά θα πρέπει να απαντήσω ε, για αυτό το θέμα το πολύ ευαίσθητο της εκμετάλλευσης ε, των ε, πετρελαϊκών αποθεμάτων στην Αδριατική θάλασσα. Να σας πω λοιπόν το εξής. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει ε, να τα λέμε απ' έξω απ' έξω. Θα πρέπει να μιλήσουμε καθαρά εάν μιλάμε για διαδικασίες εξόρυξης πετρελαίου στην Αδριατική. μιλήσμονούμε πάντω πάντως ότι οι φίλοι από την Ιταλία ήδη ε, κάνουν τέτοιου είδους ε, κινήσεις στην Αδριατική εδώ και μια δεκαετία και επομένως είναι σημαντικό ε, ε, ερώτημα γιατί δεν θα πρέπει άλλες χώρες να κάνουν τέτοιου είδους ε, προσπάθειες εξόριξης στην Αδριατική π.χ. η Κροατία. Ε, βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι εξορίξεις είναι πολύ κοντά σε τουριστικές περιοχές της Κροατίας και μη λησμονούμε ότι ο τουρισμός είναι ή ε, ε, συνώνυμος με την επιβίωση αυτών των περιοχών ε, όσο και η αλληλεία βέβαια σε πολλές περιπτώσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να σταλούν πολύ ισχυρά μηνύματα όσον αφορά την εξόριξη πετρελαίου και τις διαδικασίες αυτές στην Αδριατική η εξόριξη, η εκμετάλλευση πετρελαϊκών ε, αποθεμάτων είναι ένα θέμα, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, βοηθήσουμε και την ανάπτυξη της οικονομίας των περιοχών. Αλλά λέω θα πρέπει παρόλα αυτά σχετικά με το θέμα αυτό να στείλουμε κάποια πολύ ισχυρά μηνύματα. Ε, αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ για ό,τι μας είπατε. Ευχαριστώ για τη συμβολή σας στη συζήτηση. Η γραμματεία της Επιτροπής μας ε, θα στείλει ως ονούπο προσκλήσεις ε, στα ενδιαφερόμενα, στα εμπλεκόμενα μέλη έτσι ώστε να συνεργαστούμε και να συνεδριάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γιάκοφτσίτσε. Θα περιμένουμε το προσχέδιο της έκθεσής σας για τον μήνα Ιούνιο, σε κανένα μήνα δηλαδή, έτσι ώστε να κάνουμε την συζήτηση έχοντας πλέον το έγγραφο. Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Η Επιτροπή Μεταφορών του Κοινοβουλίου εκπονεί ε, έκθεση πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και εμείς ως Επιτροπή ε, συμμετέχουμε, συμβάλλουμε με μια γνωμοδότηση. Στο πακέτο για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα η Κομισιόν προσπαθεί να προωθήσει συνολικά το θέμα αυτό. Αυτό ήταν και ο στόχος άλλωστε της δημιουργίας αυτού του πακέτου. Ε, καταδεικνύει μοντέλο συνεργασίας, βέλτιστες πρακτικές, ε, καινοτομίες και χρήσεις της κοινοτομίας ε, μέσα στα πλαίσια αυτού, αυτής της δέσμης. Σήμερα ο συντάκτης της γνωμοδότησης, ο κύριος Ραμόν Λουίς Βαρκάθελ, θα μας παρουσιάσει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΡΕΤΖΙ για την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ε, επ' αυτής δηλαδή της εκτέσεως πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαρκάθελ. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ξέρετε κι εσείς πως το θέμα αυτής της κινητικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και κυρίως για την ανάκαμψη την οικονομική της Ευρώπης για να πετύχουμε και τους στόχους μας ε, τους, για το περιβάλλον, για τις καθαρές πόλεις. Η κρίση στην Ουκρανία και η οικονομική κρίση στην Ευρώπη μας τοποθετούν σε ένα πλαίσιο όπου τελικά είναι αναπόφευκτο να έχουμε ενεργειακή εξάρτηση, ε, να έχουμε ε, ανάγκη να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και να έχουμε και ένα, μία ακόμα ανάγκη να αυτονομηθούμε παρόλη την εξάρτηση αυτή ενεργειακά. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να το κατακτήσουμε αυτό, να έχουμε πιο καθαρές πόλεις, και παράλληλα να αναπτύξουμε μια πιο καινοτόμο οικονομία η οποία θα δώσει θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές στην Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν μπορούμε να το κατακτήσουμε και στη γνωμοδότησή μου βασίζουμε σε τρία σημεία. Καταρχήν, αυτή η βιώσιμη προσπάθεια μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ε, ε, τα κονδύλια από το ΕΚΠΑ ε, κάνοντας μια αναλύση πολιτική και ποσοτική για το πώς έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα η πολιτική συνοχής ε, για την κινητικότητα, την αστυνομική κινητικότητα, χρησιμοποιώντας τα κονδύλια που ήταν πάντα διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις να αναπτυχθούν με τον ίδιο τρόπο και να έχουν τέτοια σχέδια βιώσιμα σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα αστικά περιβάλλοντα, για να δούμε πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Να στηρίξουμε λοιπόν τις πόλεις και τις περιφέρειες έτσι ώστε να εφαρμόσουν αυτά τα σχέδια της αστικής βιώσιμης κινητικότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συντονίσει τα εργαλεία τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα και να μας ε, καταθέσει τα εγχειρίδια τα οποία μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα κατευθύνουν και τις περιφερειακές αρχές και τις πόλεις μας που είναι οι βασικοί παίκτες, οι πιο υπεύθυνοι παίκτες τη στιγμή της εφαρμογής αυτών των σχεδίων. Τέλος, θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται με τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτήσει το πακέτο Juncker. Πώς θα συντονιστούμε σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες για το πώς μπορούμε να μετακινούμαστε στις πόλεις μας με ένα βιώσιμο τρόπο. Αυτές είναι οι γενικές γραμμές ε, της ε, γνωμοδότησης που συντάσσω και θα ακούσω με μεγάλη χαρά όλες τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που έχετε να κάνετε. Πιστεύω πως οι παρατηρήσεις σας και οι τροπολογίες που θα καταθέσετε μπορεί να με βοηθήσουν να βελτιώσουμε το κείμενο έτσι ώστε να έχει το ιδιαίτερο βάρος που χρειάζεται στην Επιτροπή Μεταφορών. Αυτά λοιπόν. Και σας ευχαριστώ που μου δώσετε το ρόλο. And now give the floor. Ευχαριστώ, κύριε Βαλκάρσελ. Περνάμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές. Κυρία Κρέλεξ, ονοματός κυρία Σμόλκοβα. Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. κυρία Σμόλκοβα που μου ζήτησε να μεταφέρω κάποιες παρατηρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Για εμάς είναι σαφές πως η κινητικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τους κατοίκους των πόλεων αλλά σχετίζεται και με άλλες εξελίξεις. Μιλήσατε για την οικονομία της ΑΠΕ, την κλιματική αλλαγή, βεβαίω γιατί η μετακίνηση είναι σημαντικό κομμάτι του διοξιδίου του άνθρακα που εκλείεται στην ατμόσφαιρα και άρα χρειάζονται έξυπνες και βιώσιμες λύσεις. Οι πόλεις ήδη έχουν συχνά μεγάλο πρόβλημα με την κίνηση. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα και απαιτείται από τις πόλεις να αναπτύξουν νέα μοντέλα και η κυρία Σμόλκοβα, η σκιώδης εισηγήτρια, θα ήθελε να πούμε πως κατά τον προγραμματισμό τέτοιων λύσεων πάντα καλό είναι να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι όταν φτιάχνουμε δρόμους π.χ. και οι PC και οι ποδηλάτες. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την αηφορία. Η κυρία Σμόλκοβα χαιρετίζει την ευρωπαϊκή αυτή πλατφόρμα που προτείνει η Κομισιόν και θα ήθελε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία για έξυπνα συστήματα μεταφορών και αποδίδει μεγάλη σημασία στην διαπίστωση πως υπάρχουν κάποιες έξυπνες πόλεις με έξυπνα συστήματα μεταφορών και θα μας βοηθούσαν νομίζω για να δημιουργηθεί μια υποδομή στις πόλεις η οποία θα είναι ανθεκτική ε, για το μέλλον και βεβαίως θα ήθελε να υποστηρίξει και τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος σκιώδης εισηγητής, ε, η κυρία Βάνερ, όχι. Ο κύριος Πορέμπα δεν είναι εδώ. Οπότε, ο κύριος Γιώαντ έχει το λόγο. Κύριε Γιάκοπτιτς, θέλετε να μιλήσετε. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω εξ ονόματος ε, της ομάδας μας, της Άλτε, θα είμαι πολύ σύντομος. Συμφωνώ με όσους ήδη μίλησαν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα ήθελα μόνο να πω τα εξής. Όταν μιλάμε για την ε, κινητικότητα εντός των πόλεων, θεωρώ πως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε καθαρά καύσιμα και οχήματα και θεωρώ πως ο δημόσιος ε, τομέας εντός των πόλεων να χρησιμοποιεί πρώτος αποτελεσματικά την ενέργεια. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω, το οποίο δεν αναφέρθηκε και πρέπει να συμπεριληφθεί. Είναι κάτι συγκεκριμένο και σημαντικό. Είναι η κινητικότητα μεταξύ των πόλεων. Όταν μιλάμε για πόλεις οι οποίες κοντά στα σύνορα είναι μεθοριακές αλλά κατ' ουσίαν είναι μία πόλη όπως η Νόβα Γκόριτσα ας πούμε μέρος της οποίας είναι στη Σλοβενία και άλλο κομμάτι της είναι στην Ιταλία και πρόκειται για μία πόλη και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα στην Ευρώπη και θεωρώ πως πρέπει να μπει στην έκθεση. Και νομίζω πως είναι μια καλή ιδέα να υποστηρίξουμε την διασυνοριακή κινητικότητα και πρέπει να μπει στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ο Ζουλό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη γνωμοδότηση και να κάνω μία χωροταξική παρατήρηση. Επειδή είμαι δήμαρχος μιας μέσου μεγέθους πόλης, να σας πω πως είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε πως για την αστική κινητικότητα θα πρέπει να γνωρίζουμε πως οι πόλεις είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, ανεξάρτητα από το μέγεθος. Εγώ είμαι δήμαρχος σε μια πόλη 15.000 κατοίκων και είναι τελείως διαφορετικές οι λύσεις που μπορούμε να προκρίνουμε εμείς από ότι τι θα από ότι ε, θα πρότεινε κανείς για το Παρίσι. Επειδή οι λύσεις δεν είναι οι ίδιες, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκεί που θα δώσει προτιθέμενη αξία, που είναι οι μεγάλες μεγαλοπόλεις, θα πρέπει να μιλήσει για διάφορες ε, αστικές ζώνες και να πει πως υπάρχουν ε, ε, και κάποιες πόλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσαν να συντονιστούν μεταξύ τους και να προετοιμάσουν τα δικά τους προγράμματα για την βιώσιμη αστική κινητικότητα, πόλεις 10, 15, 20 χιλιάδων κατοίκων και να είναι και επιλέξιμες για κάποια προγράμματα έτσι ώστε να ενισχύσουμε την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Να δούμε τι σημαίνει αυτό για μας τι μιλάμε για ε, τα τραμ, για τα ε, ποδήλατα, για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, ε, για κάποιους κόμμους υδροδρομικούς, οδικούς. Τι ακριβώς σημαίνει. Ξέρετε τι συμβαίνει χωροταξικά. Δεν έχουμε μόνο μεγαλοπόλεις, έχουμε και μέσου μεγέθους πόλεις και αυτές θα πρέπει τη σειρά τους να ενθαρρυνθούν. Thank you. Thank you, No. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δεμάτου. Α, θέλετε Το θέμα το οποίο ασχολείται ο συνάδελφος της βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι ένα θέμα ιδιαίτερα προσφυλές σε όλους μας. Υπάρχουν πολλά στοιχεία σημαντικά στην έκθεση, κυρίως δε ότι ε, τα σχετικά ταμεία θα πρέπει να συμβάλλουν ε, στην εκπόνηση ε, επιχειρησιακών προγραμμάτων όπου η αστική κινητικότητα θα γίνεται μέσα από καθαρές μεταφορές και από μεταφορές ε, οι οποίες ε, ε, δεν θα δημιουργούν προμόλυνση. Ας πούμε ανανεώσιμες πηγές, zero emission transport κτλ. Ε, η Κομισιόν στα πλαίσια της δικιά της ενδιάμεσης ε, αναθεώρησης ε, της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων και επενδυτικών ταμείων είναι καλό που γίνεται αυτή η γενικότερη συζήτηση έτσι ώστε να υπάρξει βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ενδεχομένως πολλές χώρες να κρύψουν πίσω από αυτό το γενικότερο θέμα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας κάποια θέματα τα οποία δεν θα είναι ούτε αποτελεσματικά, ούτε βιώσιμα, ούτε πράσινα. Δεν αναφέρομαι βέβαια σε όλες τις χώρες προς Θεού. Αλλά ε, ξέρουμε ότι και στην, ε, ε, στη δικιά μου χώρα, σε περιπτώσεις όπως το ΤΑΒΕ ή η ΕΞΠΟ, το τρένο η ταχύτητας και το, η ΕΞΠΟ, βλέπουμε ότι εκεί έχει βάλει τα πλοκάμια της και το οργανωμένο έγκλημα και μάλιστα οι περιπτώσεις έχουν φτάσει ήδη στο δικαστήριο. Ε, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να αναλάβουμε την ε, τις αστικές, τους αστικούς χώρους, τους οποίους έχουμε χάσει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ε, χώρες όπως η Αυστραλία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση του κέντρου των πόλεων. Η ανάκτηση των πόλεων δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο. Ο κύριος Πορέβα είναι τώρα εδώ. Είναι σκιώδης συγητής. Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη για την ε, καθυστέρηση. αλλά ήμουν σε άλλη επιτροπή, την Επιτροπή Μεταφορών. Θα μιλήσω τώρα στη γλώσσα μου. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή, αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Νομίζω ότι έχει ε, καλύψει πολλά στοιχεία με συνεκτικό τρόπο και αρκετά ολοκληρωμένα. Μιλάμε εδώ για την βελτίωση της κινητικότητας της πόλης γιατί ξέρουμε ότι οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι υφίστανται τις αρνητικές επιπτώσεις ε, της ε, ε, κακής κινητικότητας. Πρέπει να είμαστε ορθολογιστές, να δούμε τα πράγματα με λογικό τρόπο όσον αφορά την αστική κινητικότητα. Και βεβαίως αυτή η κινητικότητα θα πρέπει να είναι βιώσιμη, πολυτροπική και φιλική προς το περιβάλλον. Ξέρουμε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής και αυτή η αλλαγή θα πρέπει να φανεί και στην αλλαγή του τρόπου μετακίνησης και της, ε, στις μεταφορές. Συχνά λέμε ότι θα πρέπει ότι ε, θα πρέπει να μειωθεί η χρήση του ιδιωτικού ε, αυτοκινήτου και να υπάρξει μετακίνηση προς ε, η μεταστροφή προς, τις, προς τα μέσα, μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Η δημιουργία λοιπόν εναλλακτικών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ε, και νομίζω ότι θα πρέπει και οι ίδιοι οι πολίτες να παίξουν ρόλο, να πάρουν δηλαδή οι ίδιοι αποφάσεις σχετικά ε, με το πώς θέλουν να είναι οι πόλοι τους και πώς θέλουν να είναι οι ε, μεταφορές τους αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, στηρίξει ε, τις ε, κινήσεις αυτές και τις αποφάσεις αυτές μέσα από την παροχή συγκεκριμένων λύσεων. Ε, δηλαδή όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε, στα κοινά προγράμματα για την βελτίωση το, της αστικής κινητικότητας που θα είναι πιο βιώσιμη και πιο καινοτόμα. Εγώ έχω κάποιες τροπολογίες τις οποίες θα υποβάλω και οι οποίες πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση που μόλις ανέφερα. Θα συνεργαστώ βέβαια με τον εισηγητή, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Χέντμαν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να τονίσω πως το έγγραφο είναι πραγματικά εξαιρετικό. Καλύπτει μια σειρά από θέματα τα οποία συζητάμε και σε αυτή την Επιτροπή και σε άλλες και θα μπορούσα να συνεχίσω απευθύνοντας όλο και περισσότερο συγχαρητήρια, αλλά πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι πως ο εισηγητής αναφέρεται σε μια πρωτοβουλία η οποία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, και αυτό θα αποτελέσει τμήμα της όλης διαδικασίας για τη βιώσιμη πολιτική μεταφορών μέσα στις πόλη μας. Μιλάμε για το περιβάλλον, για τα καθαρά καύσιμα και για ένα βαθμό εναρμόνισης. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω στα σχόλια που έκαναν οι προλαλήσαντες και να τονίσω πως οι βιώσιμες η βιώσιμη αστική κινητικότητα μπορεί και αυτή με τη σειρά τη να συνεισφέρει σε μεγαλύτερη οδική ασφάλεια. Και νομίζω ότι αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό να καταγραφεί. Με καινοτόμε λύσεις οι αστικές περιοχές θα μπορούσαν να γίνουν πιο ελκυστικές, για παράδειγμα. Και αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να συνεισφέρει σε βελτιωμένη ποιότητα ζωής και σε μια πιο εύκολη ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματική ζωής, να περνάει κανείς λιγότερο χρόνο στις συγκοινωνίες, έτσι ή στην κίνηση, να μπορεί να περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του και βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με το πόσο κοστίζουν οι αστικές συγκοινωνίες ειδικά για τα άτομα με αναπηρίες. Για το λόγο αυτό εγώ θα υποβάλω και τη σχετική τροπολογία. Ή τροπολογίες. Επαναλαμβάνω πως οι τροπολογίες αυτές είναι για μια άριστη γνωμοδότηση. Ο κύριος Βανλίσερο είναι ο επόμενος μιλητής Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την προσέγγιση της ε, έκθεσης αυτής της γνωμοδότησης και βεβαίω την σχέση που υπάρχει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις έξινες πόλεις και το σχέδιο Juncker. Να κάνω τώρα κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις. Εγώ δεν βλέπω τη λέξη ποδήλατο εδώ μέσα. Δεν βλέπω το ποδήλατο. Έχουμε πολύ καλή δημόσια συγκοινωνία, μπαίνει μέσα ο κόσμος και μετά βγαίνει και τι κάνει, πάλι ο κόσμος παραμένει παχουλός έτσι γιατί δεν ασκείται. Να, να πω λοιπόν την Ολλανδική άποψη, την Ολλανδική σκοπιά. Πάει κανείς στο σταθμό του τρένου και έχει χιλιάδες ποδήλατα α, παρκαρισμένα απ' έξω και μπαίνει στο τρένο. Έτσι και έτσι θα απομακρυνθούμε και από τα ορυκτά κάψιμα. Αυτό νομίζω πρέπει να πούμε. Σας ευχαριστώ. Δεκτό. Νομίζω αυτό το οποίο λέτε. Μπορεί να το δοκιμάσουμε και στο κοινοβούλιο. Ο κύριος Φαν Μίλτινμπουργκ, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να καθησυχάσω τον κύριο Φανισλόη ως σκιώδης συγητής. Σας ε, διαβεβαιώ πως ε, αναφέρεται συχνά το ποδήλατο όταν μιλάμε για βιώσιμες μεταφορές. Αλλά δεν ήθελα να πω αυτό. Θεωρώ πως έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα ο εισηγητής μας. και έχουμε νομίζω αυτό το σχέδιο που λέγεται SIMS στα αγγλικά θα πρέπει όμως ε, να υπάρχει η δυνατότητα στις ε, πόλεις να χαράζουν τη δική τους πολιτική. Οι πόλεις είναι νομίζω σε θέση καλύτερα να ξέρουν πώς θα έχουν βιώσιμη αστική κινητικότητα είτε χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και την επιτυχή της επικουρικότητας. Αλλά υπάρχει και κάτι το οποίο με ανησυχεί όταν μιλάμε για την επικουρικότητα. Διαβάζουμε στην παράγραφο 8 πως ε, ζητάμε από την Κομισιόν να επεξεργαστεί διάφορους κανόνες για τη ρύθμιση στην πρόσβαση σε αστικές περιοχές ε, και διάφορα τέτοια. Τι εννοεί εδώ πέρα ο εισηγητής. Αυτά είναι η υπόθεση των πόλεων, θα έλεγα. Και δεν γίνεται να ρυθμίζονται τα πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να μας διαφωτίσει λίγο το πέρα εισηγητής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πότζεκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση αυτή είναι νομίζω πάρα πολύ ποιοτική και έχω δύο παρατηρήσεις μόνο όπως και η κυρία Σμόλκοβα θα συμφωνούσα και εγώ πως καλό θα ήταν να συμπεριλάβουμε μία απέτηση σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να περιλαμβάνει και εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών αρχών. Στο βαθμό που μπορούν να εκπροσωπούν περιφέρειες και πόλεις διαφορετικού μεγέθους. Έτσι, έχουμε μια εγγύηση ότι οι πλατφόρμες αυτές ε, θα έχουν τα αποτελέσματα που χρειάζονται οι πόλεις. Και το ίδιο ισχύει και για τις διάφορες ομάδες ε, συμφερόντων, όπως αυτές που προωθούν την ποδηλασία. Πρέπει και αυτοί να ακούγονται και να επισημάνω ένα παράδοξο εδώ πέρα που προκύπτει από την έκθεση. Θέλουμε περισσότερους πεζούς, περισσότερους πόδιλάτες, αλλά ταυτόχρονα αυτό σημαίνει περισσότερα ατυχήματα, τραυματίες. Πρέπει να γίνει λοιπόν κάποια μελέτη που θα δείχνει τις αιτίες των ατυχημάτων και το πώς θα μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων. Μεταξύ των ποδηλατών όπως ο κύριος Φαν Ρόι. Νομίζω πως οι λύσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή πλησιάζουν στα όρια τους. Πρέπει να είμαστε πιο καινοτόμοι. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι η εξής. Το πρόβλημα είναι οι μεταφορικές δυνατότητες των ε, πόλεων. Δημιουργούνται διάφορα προβλήματα όπως η ρήπανση κτλ. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε σε παρακαπτήριες ε, για να μην διέρχεται η κυκλοφορία μέσα από την πόλη θα πρέπει ίσως να απευθύνουμε έκκληση στις πόλεις να επενδύσουν σε τέτοιες υποδομές. Για να μην έχουμε τόση κίνηση στις πόλεις. Και να απευθύνουμε έκκληση στην Κομισιόν, γιατί αυτά τα έργα κοστίζουν πολύ. Και βέβαια αυτό αφορά εξίσου και το σημείο 7 και 8 του σχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τώρα, κύριε Βαλκαρσέλ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε σε ερωτήσεις ή να κάνετε κάποιες ε, παρατηρήσεις. I'm sorry, Mr. Συγχωρείτε. Ξέχασα την Κομισιόν. Δεν το συγγνώμη. Δίνω τον λόγο στον κύριο Λίντμπεργκ από τη Γενική Διεύθυνση μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ όσους ασχολήθηκαν με την γνωμοδότηση, τον συντάκτη και τους σκιώδης και να σας διαβεβαιώσω πως όλες οι προτάσεις που κάνετε είναι πολύ σχετικές με το αντικείμενο. Όπως έχουμε υπογραμμίσει και εμείς σε σχέση με την πολιτική συνοχή, στο 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχετικό πακέτο, ακολουθώντας μια χαλαρή πολιτική προσέγγιση για την κοινή δράση σε ε, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στις μεταφορές. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να μεταφράσουμε τα λόγια σε πράξη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια απέτηση για τέτοιου είδους βιώσιμη πολιτική, αλλά έχει γίνει μια σαφέστατη σύσταση προς τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα ταμεία συνοχής έτσι ώστε να αναπτύξουν τέτοιου είδους σχέδια για βιώσιμες αστικές μετακινήσεις. Στα επιχειρησιακά προγράμματα αρκετών χωρών ήδη έχει τοποθετηθεί αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Να αναφερθώ επίσης σε μια πλατφόρμα την πλατφόρμα για τις ε, βιώσιμες αυτές μετακινήσεις που αποτελούν ένα εκ των όνου εργαλείο και πρέπει να σας πω πως το παρατηρητήριο και ο ισότοπός του για το θέμα αυτό των βιώσιμων αστικών μετακινήσεων είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να το κοιτάξετε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε. Ο κύριος Βαλκασέρ, το λέει επόμενος ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω το τέλος μάλλον. Θα απαντήσω στον κύριο Μίλτερμπουχ για το ποιο είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Πόλεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για κατευθυντήριε γραμμές με γενικό τρόπο. Είναι οι περιφερειέ οι ίδιε και κυρίω οι πόλεις οι οποίες είναι υπεύθυνε για το θέμα αυτό και θα πρέπει τα σχέδια αυτά της κινητικότητας να τα προετοιμάσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το μόνο που κάνει είναι να παρουσιάζει γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Ο κύριος Βανίστελο, κοιτάξτε, εγώ Ολλανδός δεν είμαι, αλλά βέβαια συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας. Γιατί αυτό που προτείνετε βασίζεται σε ένα πολύ στέρεο επιχείρημα. Δεν είναι τυχαίο όταν, το τι συμβαίνει, ε, το να εισάγουμε το ποδήλατο ε, στην ε, γενικότερη έννοια της αστικής κινητικότητας. Νομίζω πολύ σωστά το θίξατε και τελικά, εάν δείτε τις προτάσεις που κάνουμε που είναι 13 σημεία, θα δείτε πως πολλές φορές έχουμε συμπεριλάβει στοιχεία τα οποία συζητήσαμε εδώ κάποια άλλα όχι, γιατί υπάρχουν περιορισμοί. Όχι μόνο χρονικοί που και εκεί υπάρχουν, αλλά και ε, όγκο Πάντως αυτό που προτείνεται είναι μια πολύ καλή ιδέα, πολύ ενδιαφέρουσα και σίγουρα πολλά από αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε για να εμπλουτίσουμε το έγγραφο αυτό, σίγουρα. Και να σας πω πως κάτι είναι για μένα σαφές το οποίο σας αποτελεί και τον πυρήνα του θέματος. Η πράσινη οικονομία δεν είναι ένας όρος ο οποίος εύκολα γίνεται αποδεκτός. Η βιωσιμότητα και ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι έννοιες συμβατές με την οικονομική ανάπτυξη. Και νομίζω ότι έχει αποδειχτεί αυτό. η ανάπτυξη και η οικονομία έχουν ένα πυλώνα πάνω στο οποίο βασίζονται που είναι ο σεβασμός προς το περιβάλλον. Δεν υπάρχει λοιπόν οποιοδήποτε ασύμβατο ή οτιδήποτε σχετικό. Νομίζω ότι το ένα έχει ανάγκη το άλλο. Είναι αλληλένδετα και τα όσα είπατε για την οδική ασφάλεια ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Όπως επίσης για το πώς μπορεί κανείς να συμφιλειώσει την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή. Παρόλο που αυτό μοιάζει ξένα με τη γνωμοδότησή μα, η κινητικότητα, η βιώσιμη ε, κινητικότητα σίγουρα σχετίζεται και με αυτά τα δύο σχόλια. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσες λοιπόν οι παρεμβάσεις σας και γι' αυτό σας ευχαριστώ ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους συνεισέφεραν στη συζήτηση, γιατί πραγματικά εμπλουτίζουν το κείμενο, το είπα και στην αρχή της παρέμβασής μου της πρώτης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Προτείνω για τις τροπολογίες Τετάρτη 13 Μαΐου το μεσημέρι, 13 Μαΐου, λήξη της προθεσμίας υποβολής τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Και τώρα, να σας πω ότι ολοκληρώσαμε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως για σήμερα και θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών αλλά και κλεισμένων των θυρών. Παρακαλώ λοιπόν να παραμείνουν μόνο οι συντονιστές. οι τους.